Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουν έρθει όλοι, αλλά ας αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Όλοι καλωσορίσατε. Και το πρώτο θέμα σήμερα στη διάταξη είναι η έγκριση αυτής Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι κάπως ίσως πρέπει να αλλάξουμε ε, τα, τα, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις τη σειρά δηλαδή των θεμάτων γιατί πρέπει να φύγει ο συνάδελφος Μποσινάρου αλλά να ακούσουμε πριν φύγει τι έγινε με τις διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Συνοχής ε, και μετά να πάμε στο, ε, στο, στο, στα υπόλοιπα θέματα. Αυτά ε, γιατί πέραν τούτων δεν έχουμε άλλο έτοιμα αλλαγή στην ημερησία διάταξη. Ε, υπάρχει μετάδοση στο ίντερνετ της ε, και ε, όπως συνήθως ε, θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμα της ε, συνεδρίασης, το ορολόγιο, μόνο θεωρητικό είναι. Οπότε μπορεί να το έχετε υπόψη σας αυτό γιατί μπορεί να πάσα στιγμή να αλλάξει και εδώ ξέρετε κάτι άλλο τώρα έχουμε την έγκριση των πρακτικών των ε, συνεδριάσεων 18-19 Μαρτίου και 22-23 Απριλίου και ως συνήθως τα πρακτικά έχουν ε, διανεμηθεί και ε, δεν υπάρχει κάποια ένσταση τα πρακτικά αυτά θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Θέλω να σας κάνω μια ανακοίνωση, να σας παρουσιάσω το πώς βλέπω τη διαδικασία σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, σε σχέση με τη δουλειά μας. Βέβαια, ε, για να αξίζει τον κόπο θα ήθελα να είναι κόσμος να τα ακούσει, γι' αυτό και θα σας τα πω λίγο αργότερα που θα έχουν έρθει περισσότεροι συνάδελφοι. Τώρα όσον αφορά το σημείο υπαριθμών 4 της μιας διατάξεως. Η εφαρμογή της Αττικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία 2010-2012. Εδώ θα συζητήσουμε το σχέδιο κειμένου. Έχουμε εδώ τη συντάκτρια, την κυρία Μαρτίνα Άντερσον. Σας δίνω τον λόγο. Πρόκειται για τις συνέπειες Τη οικονομική κρίσης για την νεολαία. Δεν μπορούσαν ε, να δουλέψουν όπως πριν, δεν μπορούσαν να κάνουν τις, ε, τις ε, σπουδές τους. Έχουμε 6 εκατομμύρια ήδη ε, άνεργους, 50% ή παραπάνω στην Ισπανία και πολύ σε άλλες χώρες. Οπότε έτσι όπως πάμε θα αυξηθούν αυτοί και πάρα πολλοί βουλευτές έχουν προβληματιστεί και γι' αυτό και εγώ θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την κινητικότητα, τι θα γίνει με τη μετανάστευση, γιατί αυτά μπορούν να βοηθήσουν. Ιδίω όσον αφορά την μετανάστευση στην Ισλανδία, έχουμε κάποιε μακρόπνες ε, δυσκολίε, ε, πολλέ κοινότητε έχουν πληγεί και, ε, και σήμερα κιόλα μπορεί να διαβάσετε ρεπορτάζ στον τύπο που αναφέρουν το τι επιπτώσει έχουμε σε όλη την Ισλανδία σε, σε κομμοπόλεις, σε πόλεις και του κυρίου Άντζελη έχουμε μία τροπολογία τη θεωρώ πάρα πολύ θετική το 2011 σύμφωνα με την Κεντρική Στατική Υπηρεσία πάνω από 80.000 μετανάστευσαν από το, την Νότια Ιρλανδία και το 2012 διαπιστώνουμε ότι η μετανάστευση αυξήθηκε και πήγε στις 87.000 και 47.000 και μισό από αυτούς ε, ήταν Ιρλανδοί πολίτες, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό για τις κοινότητες και άλλοι για τις οικογένειες. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το κοινωνικό οικονομικό κόστος, να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, οι επιπτώσεις για τις κοινότητες σε όλα τα κράτη-μέλη. Πολλοί ευρωβουλευτές έχουν ε, επισημάνει τα προβλήματα. Τι γίνεται λοιπόν στη χώρα εκάστοτε. Συμφωνώ με την τροπολογία 1α σε σχέση με το ότι εάν δεν κάνουμε κάτι για την ε, ανεργία ε, τότε αυτό θα μειώσει την εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα πληγεί η δημοκρατία αυτά λέει η κυρία Σάντσες Σμιτ στην ε, τροπολογία της θα πρέπει κάτι να γίνει για την μακροπρόθεσμη ανεργία θα πρέπει επομένως να υπάρξουν πόροι που να βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και επίσης σε μια άλλη τροπολογία λέμε ότι ο ILO ε, έχει εγκρίνει μια προκοδόση 21 δισεκατομμύρια όμως ε, μόνο 6 από αυτά τα δις έχουν διατηρηθεί για σήμερα. 6 δις δεν αρκούν εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μακροπρόθεσμης ενεργείας. Επίσης θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή, να φέρουμε κοντά μας τους νέους, να τους δώσουμε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα των εγγύσεων και να έρθουμε σε επαφή με το European Youth Forum, με τους άλλους φορείς των νέων. Ε, εγώ ήρθα σε επαφή με το φορέα αυτό στην Βορειοελλανδία και είπαν ε, το πόσο έχουν πληγεί οι νέοι κατά την κρίση, χρειάζονται το Ταμείο Εγγύησης και στις 7 έκτου πρόκειται να οργανώσω μια εκδήλωση στην Ιρλανδία και ε, θα έρθουν εκπρόσωποι των νέων από όλη τη χώρα. Θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και ελπίζουμε έτσι να ασκήσουμε κάποια επίδραση, επιρροή ε, προς ε, ευρωβουλευτές, γενικά προς τα θεσμικά όργανα κάτι να κάνουν. Ευχαριστώ όλους όσοι ανεπλάγησαν στην ε, σύνταξη αυτού του κειμένου, κυρίως τους ε, ευρωβουλευτές, συναδέλφους που πρότειναν κάποιες τροπολογίες που είναι πάρα πολύ χρήσιμες και τελικά ελπίζω ότι θα έχουμε ε, μια στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματική ούτω ώστε να αποτελεσματική η αντιμετώπιση της ενέργειας των νέων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα έχουμε τους όλους εισηγητές. Ο συντονιστής του ΕΛΚ, Φανής Ευχαριστώ πολύ. Στείλαμε έναν από τους νεότερους εκεί, αλλά τώρα δεν μπορεί να είναι παρόν, οπότε θα αναλάβω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι να υπάρχει ευθυγράμμιση με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, όταν μιλάμε για αυτές τις πρωτοβουλίες. Και το πιο σημαντικό βέβαια είναι η ευαισθητοποίηση σε αποκεντρωμένο επίπεδο, ότι εκεί πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Εκεί αρχίζει όλη η αλυσίδα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκεί ακουμπάμε την πραγματική κατάσταση και βλέπουμε πώς θα ε, συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την ανάπτυξη στην αγορά εργασίας και τον αριθμό των νέων που θέλουν να βρουν δουλειά. Γιατί όλα αυτά γίνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι σημαντικό αυτό. Δεύτερον, αν δείτε τα δημογραφικά, βλέπουμε μια στασιμότητα λόγω της οικονομίας, λόγω της ε, ε κρίσης Έχουμε μια προσωρινή κατάσταση, γιατί αν δείτε την εξέλιξη των δημογραφικών στην Ευρώπη σε 10-15 χρόνια, σε πολλά μέρη της Ευρώπης, θα έχουμε έλλειψη νέων εξοπλισμένων ανθρώπων. Και αν δείτε και μακροπρόθεσμα τους ηλικιωμένους που θα θέλουν φροντίδα, βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα και έλλειψης και στην υγεία και στις υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους. Οπότε είναι καλή η επένδυση να κρατήσουμε ε, ζωντανές τις θέσεις εργασίας και τις υπηρεσίες πρόθεσμα. Η επένδυση σήμερα στους νέους σημαίνει ότι εξοπλίζουμε νέους για την αγορά εργασίας, στις υπηρεσίες, την πραγματική οικονομία και όπως είπα και θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας που χρειάζονται. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί τώρα εμείς να δώσουμε στους νέους την δυνατότητα να μπουν στην αγορά εργασίας, να αποκτήσουν εμπειρία και να μην χάσουμε αυτούς τους ανθρώπους από την αγορά εργασίας. Αυτό ήθελα να πω μακροπρόθεσμα θα αλλάξει η κατάσταση, δεν θα είναι όπως είναι τώρα, οπότε αξίζει να επενδύσουμε στους νέους. Δεύτερον, το ποσό βέβαια μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσό, αλλά αν δεν έχουμε πολλά λεφτά πρέπει αυτά που έχουμε να τα δαπανίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να κάνουμε περισσότερα με τα ίδια λεφτά, όχι κατά ανάγκη λιγότερα, με λιγότερα λεφτά περισσότερα πράγματα. Υπάρχει ένας ε, ε, νόμος των επενδύσεων κάθε και ε, αυτό ε, δεν μπορεί να ισχύσει παντού αλλά θα πρέπει να δουλεύουμε με ολοκληρωμένο τρόπο και να επενδύουμε καλύτερα. Έχουμε το κοινωνικό ταμείο πολλές δράσεις θα διοργανωθούν εκεί στο, με το νέο χρηματοδοτικό μέσο μαζί με τα παλιά και χαίρομαι διότι και από το ΕΤΠΑ και από το Κοινωνικό Ταμείο ε, υπάρχουν λεφτά για να επενδύσουμε στις υποδομές και να φτιάξουμε καλύτερα σχολεία όπου χρειάζεται, για παράδειγμα. Ίσως χρειάζονται περισσότερα χρήματα, αλλά πρέπει να είναι στοχευμένη η χρήση των χρημάτων μέσα στα πλαίσια των ταμείων. Ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει δυνατότητα να προβλέψουμε στον επόμενο προϋπολογισμό ή των επομένων ετών τους προϋπολογισμούς να προβλέψουμε περισσότερα κονδύλια. Ο κύριος Λεχάν θέλει να τονίσει την επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν συγκρίνουμε την Ευρώπη με τις Ηνωμένε Πολιτείες για παράδειγμα αλλά επισκεφθήκαμε και την Κορέα επίσης και είδαμε πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα τους εκεί. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τα αποτελέσματά μας στην ε, ε, οικονομία με τις νέες, στην τεχνολογία των πληροφοριών. Πρέπει να δημιουργήσουμε περιβάλλον για όλα αυτά, να δώσουμε κίνητρα. Τώρα βλέπω, είναι συνδεδεμένος εδώ ο παρακαθήμενός μου. Ε, αν υπάρχει δικτύωση μπορούμε να έχουμε συνεργασία ευρύτερη. Δεν χρειάζεται δηλαδή αστικό περιβάλλον μιας πόλης για να ε, αναλάβουμε δημιουργική δράση στη νέα οικονομία. Και τώρα ε, η, ε, μια, στις πέντε θέσεις εργασίας θα έχουν σχέση με το ίντερνετ. Αυτά μπορούν να γίνουν παντού στην Ευρώπη αν μπουν σωστά οι βάσεις, δημιουργηθεί δηλαδή το κατάλληλο περιβάλλον. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που έχει να πει η ομάδα μας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα γιατί το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, τεράστια η πρόκληση, αλλά αν δούμε με οριζοντα 10-15 ετών μπορούμε να έχουμε αλλαγή αυτής της προσωρινής κατάστασης και θα χρειαστούμε ε, καλά καταρτισμένους, με κίνητρα νέους. Χρειαζόμαστε όλους τους νέους στην Ευρώπη. Τους χρειάζεται η κοινωνία. Και δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για χαμένη γενιά, δεν θα γίνει σόνι και καλά έτσι. Θα τους οδηγήσουμε κάπου. Εκεί όπου υπάρχει παιδεία, εκεί που υπάρχουν θέσεις εργασίας, μόνο έτσι γίνεται. Ε, πήγα πρόσφατα στο Δουβλίνο και άκουσα και τον Υπουργό Παιδείας σας και είπε ότι ε, δημιούργησαν πέντε ε, ενιαία κέντρα στην Ιρλανδία. Ήταν περήφανος για αυτά που συνδυάζουν, μεταξύ, συνδυάζουν τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τις τρεις όχι μόνο πανεπιστημική, αλλά τριτοβάθμια, για να εξοπλιστούν καλά για τις αυριανές θέσεις εργασίας οι νέοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Ε, επενδύσεις λοιπόν σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο πόλεων είναι πολύ σημαντικό ε, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά μας μέσα. Ευχαριστώ πολύ Λάμπερτ και η κυρία Βασιλίσσα Βιολίτσα Δαντσίλα για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρώτη περίοδο 2010-2014 καταδεικνύει το ρόλο της νεολαίας, της δράσης που προτείνει η Επιτροπή, καθώς και για πολυδιάστατες δράσεις υπέρ των νέων. Επειδή πρόκειται για ένα πολυτομιακό μέσο και αποτελεί πρότυπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για όλο τον κόσμο. Έχουν καταβάλει προσπάθειες τα κράτη-μέλη για να βρουν λύσεις ε, για τη μείωση της ανεργίας σε επίπεδο νέων και για την σύσταση ενός κύκλου κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Είναι ευεργετικό το γεγονός ότι η στρατηγική αυτή επέτρεψε στα κράτη-μέλη να παγιώσουν τις εθνικές προτεραιότητες και βοήθησε τα κράτη-μέλη στην εκπόνηση των στρατηγικών υπέρ της νεολαίας με στοχοθετημένες πράξεις και πολιτικές. Στον τομέα ε, ιδιαίτερα της ένταξης στην αγορά εργασίας. Έτσι θεσμοθετήσαμε ορισμένες διαρθρώσεις ή εθνικούς μηχανισμούς για προγράμματα υπέρ της νεολαίας. Θεωρώ ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις και ιδιαίτερα οι νέοι εξαιτίας της κρίσης Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε άξονες δραστηριότητες, δραστηριότητας για να βοηθήσουμε τους νέους μέσα στα πλαίσια και της Ευρώπης 2020. Έτσι θα παγιώσουμε τις δράσεις κατά την επόμενη τριετία για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. ανεξάρτητα από το που ε, ε, ζουν. Είτε πρόκειται δηλαδή για μειονεκτικές περιοχές, για αστικές, αγροτικές ή οπουδήποτε αλλού κατοικούν. Πρόκειται για καινοτόμες δράσεις και επιχειρηματικές δράσεις υπέρ των νέων για να μπορέσουμε να δράξουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, ενώ στον τομέα εργασίας. Έτσι θα προσαρμόσουμε τα προγράμματα υπέρ των νέων και θα εξεύρουμε τα κατάλληλα μέσα για τη θέση σε εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Uh, thank you. I, don't see... Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον Ζανζάκ Ούτε ο ε, Βλάσακ. Ο κύριος Γκοντμάνης έχει το λόγο στη συνέχεια. έχει το λόγο. ο συνάδελφος, η συνάδελφος υπεύθυνη δεν μπορεί να παραστεί σήμερα και γι' αυτό θα ε, σχολιάσω το, μάλλον θα διαβάσω το έγγραφο που μου έδωσε και θα σας πω και μερικά δικά μου σχόλια. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να εκφαριστήσω τη Μαρτίνα Άντερσον και πιστεύω, λέει η συνάδελφος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρώπη 2020 έχει ένα βασικό στόχο, δηλαδή να μειωθεί η εγκατάλειψη του σχολείου έτσι ώστε οι νέοι να μην εγκαταλείπουν το σχολείο και τη ε, μάθηση. Τουλάχιστον να έχουμε μία βελτίωση της τάξης του 10%. Αναλύοντας όμως επιτόπια την εφαρμογή αυτού του κριτηρίου, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν καλά αποτελέσματα, δεν υπάρχει μεθοδολογία, δεν ξέρουμε πού πρέπει να επενδύσουμε γιατί το θέμα της εγκατάλειψης του σχολείου σχετίζεται με οικογενειακά ζητήματα, με την οικογενειακή κατάσταση. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά όταν ε, μας απασχολήσει και αργότερα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια κοινή προσέγγιση και μεθοδολογία για το πώς να αντιμετωπίσει το θέμα. Είναι περισσότερο κοινωνικό παρά μαθησιακό. Η κυρία Ακορίνα θεωρεί ότι σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να δούμε ε, πώς ε, οι πόλεις ε, και ε, τα περιφερειακά κέντρα θα μπορέσουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο, δηλαδή να δημιουργηθούν κέντρα νεότητας έτσι ώστε και οι μικρές περιφέρειες να μπορέσουν να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν περισσότερες ε, γνώσεις. Σε σχέση με τη μετανάστευση στην Ιρλανδία έχει δίκιο η εισηγήτρια ε, γιατί υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη μετανάστευση από τη Λετωνία και τη Λιθουανία ιδιαίτερα και ιδιαίτερα προς την χώρα σας. Ο κύριος, ε, η κυρία Πακορίνεν θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει επιπρόσθετη χρηματοδότηση και στο έρασμους να έχουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τη νεότητα. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να υπάρξει και μία ξεχωριστή γραμμή για τον προϋπολογισμό. Αυτό θα το ε, προωθήσει ε, και ο σκιώδης μας της ομάδας και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και χρηματοδότηση από τα διαφορετικά ταμεία. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα στην Ευρώπη στο τομέα της ε, επαγγελματική κατάρτισης στις ε, γερμανόφωνες χώρες είναι διαφορετικό το σύστημα σε σχέση με τις χώρες που προσχώρησαν μετά το 2004 στις γερμανόφωνες χώρες βλέπουμε ότι οι νέοι βρίσκονται σε επιχειρήσεις πολύ περισσότερο και πάρα πολύ λίγο σε κέντρα κατάρτισης ενώ στις άλλες χώρες τα, ε, οι μαθητές βρίσκονται σε, επαγγελματικά, σε σχολεία επαγγελματικής ε, κατάρτισης και όταν αφήσουν το σχολείο δεν έχουν δυνατότητα εργασίας διότι δεν γνωρίζουν τα νέα συστήματα των ε, επιχειρήσεων. Και έτσι έχουμε πολλούς αποφύτους οι οποίοι όμως δεν μπορούν να βρουν εργασία και αυτό αφορά ε, στο, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σωστές ε, δεξιότητες. Είναι δύσκολο να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα. Χρειάζονται 5 με 10 χρόνια για να ξαναχτιστεί το σύστημα και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να συμφωνήσουν υπάρχει μια βάση κατάρτισης στις επιχειρήσεις τους έτσι ώστε να υπάρχει να δοθεί μια νέα κατανομή και ιδιαίτερα ε, για, τους, ε, ε, όσους προσχώρησαν αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση είναι δύσκολη. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, συμφωνήσαμε όλοι ότι η ανεργία των νέων είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όταν δούμε όμως τα στατιστικά στοιχεία, βλέπουμε ότι στην Ολλανδία, τη Γερμανία, ο δείκτης ανεργίας μεταξύ νέων είναι κάτω από το 10%. Στη Γερμανία είναι 7,7%. Γι' αυτό νομίζω ότι οι βέλτιστες πρακτικές στα άλλα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια καλή λύση. Διαφωνώ με τον κύριο Λάμπερτ που λέει ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την αγορά εργασίας. Νομίζω ότι οι νέοι όταν αποφασίσουν ε, για τις σπουδέ τους θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το 2005 αλλά και νωρίτερα εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Πακέτο υπέρ των νέων και ορίστηκε ένα πλαίσιο κινητικότητα των νέων, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους και είχαμε και την τελευταία πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Εδώ υπάρχει υποστήριξη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, ευρώ αλλά δυστυχώς Τις θέσεις εργασίας τις δημιουργούν οι επιχειρήσεις, όχι οι πολιτικοί. Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο που να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας ή να ενθαρρύνουμε τους νέους να δημιουργούν οι ίδιοι θέσεις εργασίας ως αυτοαπασχολούμενοι. Όμως εμείς φέρουμε την ευθύνη διότι οι λύσεις μας ενέχουν πολύ υψηλό κόστος και οι επιχειρηματίες μειώνουν και την απασχόληση. Όταν δούμε τις προσφορές στην αγορά εργασίας, βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες προσφορές αφορούν εκείνους που έχουν επαγγελματική κατάρτιση. Και όσοι έχουν ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση μπορούν να βρουν θέσεις εργασίας ευκολότερα. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αφορά και τον τομέα των πολυτεχνείων, αλλά όταν δούμε τις επιλογές των νέων βλέπουμε ότι ότι ε, οι σπουδές που επιλέγουν περισσότερο ανθρωποκεντρικές, θεωρητικές δηλαδή είναι οι σπουδές τους, πολύ περισσότερο. Εμείς δίνουμε πολλά εκατομμύρια για την κατάρτιση, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει κανείς από τη δίνη της ανεργίας. Πολλές φορές απασχολούνται για έξι μήνες και στη συνέχεια γίνονται άνεργοι εκ νέου. Γι' αυτό πολλές καταρτήσεις δημιουργούνται απλώς για να δαπανηθούν χρήματα και για τίποτα άλλο. Και έτσι κατασπαταλώνται τα χρήματα του Κοινωνικού Ταμείου. Γι' αυτό θα πρέπει να διοργανώσουμε ένα φόρουμ με εκπροσώπους ανέργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ακούσουμε τη δική τους εμπειρία, να δούμε ποια εμπόδια και προσκόμματα αντιμετωπίζουν και στην συνέχεια θα τους βοηθούσαμε. Θα κλείσω το κατάλογο. Να είστε σύντομοι παρακαλώ, γιατί θα φάμε το χρόνο των άλλων εκθέσεων. Η Εμίλια Ματσόνη παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ την πρόταση αυτή που τονίζει τη σημασία της συνέχειας μεταξύ κατάρτισης και εργασίας και σε αυτό το μέτωπο θα πρέπει να συνεισφέρουμε και εμείς για να δημιουργήσουμε μέσα τα οποία πραγματικά να φτάσουν σε αυτό το στόχο. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράσω δύο σκέψεις. Ως προς τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται ότι εμείς ε, αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα σήμερα. Μιλάμε για ένα πακέτο για την νεότητα και προσπαθούμε να εξεύρουμε μέσα για αυτή τη συνέχεια και για να μην υπάρχει διάχυση ούτε στην κατάρτιση ούτε στην εργασία. Δεν βλέπουμε όμως πώς έχει η κατάσταση, η τρέχουσα κατάσταση. Θα πρέπει να μας απασχολήσει η τοποθέτηση στην αγορά εργασίας εκείνων που έχουν ακολουθήσει σχέδια κατάρτισης και σήμερα περιμένουν να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση, περιμένοντας στη συνέχεια οι νέοι αυτοί να βρουν δουλειά στην αγορά. Επίσης, η ενεργεία των νέων είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι κάτι το πολύ ανησυχητικό. Θα πρέπει να μας απασχολήσει η πολιτισμική εξέλιξη των νέων. Και γι' αυτό θα ήθελα να δούμε και το υψηλό ποσοστό γυναικών που δεν απασχολούνται. Και να δούμε τι επιπτώσεις υπάρχουν. Αυτό έχει να κάνει και με τη βία κατά των γυναικών. Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η υψηλή ανεργία έχουν μεγάλη επίπτωση επί του δραματικού αυτού φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν με αυτή την ευκαιρία να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα τα οποία σας σκιαγράφησα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Χρυσόγελος. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι ε, η ανεργία των νέων είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. Η ανεργία μεταξύ των νέων στην Ελλάδα είναι 64,2% και στην Ισπανία είναι σήμερα 56%. Άρα δεν είναι ένα φαινόμενο σαν και αυτά που ξέραμε στο παρελθόν, όπου έπρεπε να αλλάξουμε, να προσαρμόσουμε τα συστήματα εκπαίδευσης για να μπορέσουν να μπουν οι νέοι στην ε, αγορά εργασίας. Σήμερα δεν υπάρχει οικονομία στην Ελλάδα για να μπουν. Επομένω, ε, είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Έχουμε ανεργία, αλλά έχουμε και μια πλήρη κατάρρευση του παραγωγικού τομέα. Και άρα τα προβλήματα είναι διπλά. Δηλαδή θέλουμε και αναζωγόνηση οικονομίας και θέλουμε και μεταρρύθμιση και μεταβολές στο σύστημα κατάρτισης και εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να μπουν οι νέοι σε σύγχρονες ανάγκες, να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν σύγχρονα θέματα. Πολλές φορές γίνεται και ένα λάθος. Ε, προτείνονται σε περίοδους κρίσης μία επιστροφή στο παρελθόν και στο θέμα της οικονομίας, παλιοί τομείς ε, το ίδιο μοντέλο το οποίο οδηγήθηκε σε χροκοπία, αλλά και συστήματα απασχόλησης των νέων που δεν ήταν αποτελεσματικά. Δηλαδή, με ένα θέμα το οποίο έχουμε στήσει πολύ συχνά εδώ πέρα είναι το θέμα της απορροφητικότητας. Όταν λοιπόν τα προβλήματα είναι τόσο εκρηκτικά, ε, συνήθως οι κεντρικές εξουσίες αλλά και οι περιφερειακές επιστρέφουν σε μια λογική να πάνε γρήγορα χρήματα και συνήθως αυτό δεν είναι αποτελεσματικό γιατί δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός. Είναι σημαντικό λοιπόν να δημιουργηθούν ε, και καινούργιες μορφές απασχόλησης ε, και να αναζωογονηθεί η οικονομία σε καινούργιους τομείς. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν, είναι, δεν μπορούμε να λέμε στους νέους ότι μπείτε σε όποια εργασία και μπείτε με συνθήκες που μερικά χρόνια πριν θα λέγαμε ότι είναι πολύ μακρινές από τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη. Με 300 και 300 ευρώ πρέπει να δουλέψει σήμερα κάποιος στην Ελλάδα νέος, αν βρει εργασία επομένως νέους ανθρώπους μας ότι σπουδάσατε, αποκτήσατε γνώσεις ή ικανότητες και τώρα πρέπει να κάνετε δευτερεύουσες δουλειές ή ακόμα αν κάνετε και σημαντικές δουλειές η αμοιβή σας 300 300-400 ευρώ και αυτό είναι ένα ποσό το οποίο κάνει αδύνατη τη ζωή των νέων ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πάρα πολλοί νέοι, τα πιο δυναμικά μυαλά, τα πιο δημιουργικά μυαλά φεύγουν από τη χώρα και από την Ελλάδα και από την Ισπανία και από άλλες χώρες και να ζητούν εργασία στη Γερμανία, στην ε, Βρετανία ή ακόμα και πολύ μακρύτερα και έτσι χάνουμε και τις δυνάμεις εκείνες που μπορούν να βοηθήσουν στην αλλαγή της κοινωνίας, στη μεταρρύθμιση, στην αλλαγή της οικονομίας, στην κοινωνική συνοχή και στην περιφερειακή ανάπτυξη που Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Οι περιφέρειες για να μπορέσουν να προετοιμαστούν για τη νέα προγραμματική περίοδο θέλουν ανθρώπους που θα έχουν γνώση ποιε είναι οι κατευθύνσει του μέλλοντο. Μιλάμε για έξυπνη, περιεκτική, βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά αυτό μπορούν να το κατανοήσουν οι νέοι που έχουν περάσει τα πανεπιστήμια, οι νέοι που έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Αυτοί όμω οι νέοι δεν μπορούν να μπουν πια και στι περιφέρειε και σε ε, φορεί που θα προετοιμάσουν το σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Άρα λοιπόν έχουμε μία πλήρη κατάρρευση όλη τη αλυσίδα. Οι κρίκοι έχουν σπάσει και καταραίει όλο το σύστημα. Αλλά να πω μερικέ προτάσει που αναφέρονται και στην έκθεση οι περισσότερες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να βρούμε εργαλεία που γρήγορα βοηθούν τους νέους ανθρώπους να συνεχίσουν την κατάρτιση να μπουν στην απασχόληση. Το Youth Guarantee είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά εκεί που χρειάζεται δεν υπάρχουν οι πόροι. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν τέτοιε δραστηριότητε. Δεν υπάρχουν αυτοί οι πόροι. Δεν υπάρχουν και στην Ευρώπη, γιατί το ποσό που θα κατευθύσει στου νέου είναι το 0,6 του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού. Ενώ θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο και το λέγαμε εδώ πέρα ότι είναι τουλάχιστον 20 δις που χρειάζονται για τους νέους και η εκτίμηση, την ακούσαμε και άλλες φορές εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι ότι η ανεργία έχει κόστος οικονομικό 150 δις. Δηλαδή το κόστος είναι 150 δις και εμείς ως Ευρώπη επενδύουμε μόνο 6 δις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να βοηθήσουμε τους νέους να απασχοληθούν. Το δεύτερο είναι ότι χρειαζόμαστε και ευέλικτα εργαλεία. Ένα νέο άνθρωπο που θέλει να ξεκινήσει μια δραστηριότητα, άμα πάει σε μια τράπεζα, δεν πρόκειται να πάρει χρηματοδότηση. Είναι λογικό, είναι κάποιο που ξεκινάει. Και γι' αυτό χρειάζεται ευέλικτα εργαλεία. Και είναι πολύ σημαντικό σε κάθε χώρα μέλο αλλά και με ευρωπαϊκού πόρου να υπάρχουν αυτέ οι δυνατότητε για να υπάρξει μια άνθηση τη επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα σε τομεί κοινωνικού και περιβαλλοντικού, σε καινοτομία, σε, οικολογική, σε καινοτομία θα έλεγα εγώ, έτσι ώστε πράγματι οι ίδιοι οι νέοι να δημιουργήσουν θέσει εργασία μέσα από κοινωνική και περιβαλλοντική γενικότερα επιχειρηματικότητα. Γιατί ο δημόσιος τομέα δεν μπορεί να απασχολήσει πλέον και πολλοί τομεί της οικονομίας έχουν καταρρεύσει. Άρα θέλουμε νέα πράγματα. Αλλά όταν ένα νέο θέλει να ξεκινήσει κάτι, πού θα βρει του πόρους. Ούτε οι γονεί του έχουν πλέον χρήματα για να του δώσουν. Άρα πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί πλέον σε κάθε χώρα δεν υπάρχουν αυτοί οι πόροι και να δούμε τέτοια εργαλεία. Ε, είναι θετικό κατά την άποψή μου ότι ε, ο Υπουργό Οικονομικών τη Γερμανία μίλησε για κάποια παρόμοια αλλαγή στην πολιτική, την οικονομική, αλλά πρέπει σε επίπεδο ευρωπαϊκό θεσμικό να το σκεφτούμε και να δημιουργήσουμε τέτοια εργαλεία. Ευχαριστώ. Μαρία Ριγόγεν, παρακαλώ να είσαι σύντομη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Έχω τρεις παρατηρήσεις. Είναι το βασικό θέμα, το θέμα προτεραιότητας που έχουμε σήμερα. όχι, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε δουλειά σε κάποιον, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε λύσεις. Λύσεις για τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Και το πρόβλημα αυτό των νέων είναι το πιο σημαντικό. Με τις μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να έχουμε κάποιες δυναμικές πολιτικές απασχόλησης να ξαναβρούν δουλειά, να ξαναμπούν στον κόσμο, στον χώρο της δουλειάς είναι Γιατί έχουμε προσπάθειες μέσω της παιδείας που δεν ε, ε, αποδίδουν πάντα. Κοιτάξτε, στην Ισπανία δεν είναι τόσο κακή η παιδεία. Έχουμε κάποιους οι οποίοι έχουν τα προσόντα, διότι μπορεί να μην βρίσκουν δουλειά στη χώρα τους, αλλά μεταναστεύουν και βρίσκουν δουλειά. Άρα το θέμα είναι να δούμε από πλευρά οικονομίας τι θα γίνει. Το πρόβλημα για την κρίση είναι πολύ πολύ ευρύτερο από ό,τι φαίνεται. Τώρα κάτι άλλο. Ναι, συμφωνούμε ότι αυτή είναι η βασική μας πρόσκληση. βασική πρόκληση που έχουμε εδώ η πολιτική. Να μπορέσουμε στις ε, χώρες μας να, να, να προωθήσουμε την ιδέα να ενδυναμωθεί το κοινωνικό ταμείο. Και έτσι αυτοί οι νέοι που βγαίνουν από τα σχολεία, από τα πανεπιστήμια να μπορούν να βρουν δουλειά. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, κύριε Άντερσον, ε, μπορείτε να δευτερολογήσετε, αλλά παραγωνίστε και εσεί σύντομοι. Ναι, όχι, όχι, δεν, είναι δυνατόν να τα καλύψω όλα αυτά. Πάντως, ευχαριστώ όσους ε, βουλευτές έλαβαν το λόγο. Είπανε μερικά σημαντικά, ιδίω τα σχετικά που ακούσαμε για τις δημογραφικές τάσεις. Άρα, για το μέλλον θα πρέπει να Χαράξουμε προσοχή τη στρατηγική μας. Όμως θα πρέπει επίσης να δούμε τι θα κάνουμε με τα προγράμματα. Τα προγράμματα που ξεκίνησαν στο παρελθόν, να δούμε τι θα γίνει την περίοδο 2014-2020, έτσι με τα προγράμματα αυτά να κάνουμε τη διαφορά. Να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της γραφειοκρατίας για το οποίο όλοι οι φορείς παραπονούνται. Πάντως, το θέμα είναι και η επιχειρηματικότητα, πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, γιατί γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν κάποια εργαστήρια 200 παντού στον κόσμο για να, στην Ευρώπη συγγνώμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα προσόντα των νέων ε, αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Μιλάμε για αυτούς που από τα 17 ώστε να βρουν δουλειά. Ε, μιλάμε για 12 χρόνια υποχρεωτική ε, παιδείας που όταν τελειώσουν το σχολείο δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν όπως πρέπει. Άρα θα πρέπει, είπαμε και ε, στην Βόρεια Ιρλανδία να δούμε το θέμα της ε, παιδείας. Από τα 11 και μετά υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε τον 2020, έχουμε τις ε, κοινωνικοπολιτικές δραστηριότητες, οπότε θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, να δούμε τι μπορεί να γίνει μέσα από τα προγράμματα. Αυτά τα οποία τρέχουμε να τα στηρίξουμε, να τα αναβαθμίσουμε και να δοθούν έτσι οι ευκαιρίες που χρειάζονται. Τα 21 εκατομμύρια του ILO χρειάζονται, τα 6 δεν αρκούν. Θα μιλάμε για 150 εκατομμύρια που κοστίζει αυτή η ανεργία. Αυτά τα έξι είναι πενταροδεκάρες. Δεν φτάνουν. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση, όπως φάνηκε η τη σημερινή συζήτηση. Και έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση αυτής της έκθεσης ε, και να πούμε δηλαδή στον κόσμο εκεί έξω αυτά που περιμένει να ακούσει εγώ μας. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Οφείλω κάποιες εξηγήσεις για την έκθεση όταν η Επιτροπή Πολιτισμού δεν μπορούσε να περιμένει τη γνωμοδότηση γιατί ήταν λίγος ο χρόνος, θα ψηφίσουν 17 Ιουνίου εκείνη. Οπότε η μόνη εναλλακτική ήταν να σας στείλουμε τις τροπολογίες, το σχέδιο έκθεσης, χωρίς ε, τη συζήτηση, πριν από καιρό το στείλαμε, για να προλάβουμε να καταθέσουμε και τις τροπολογίες. Λάβαμε 28, η συζήτηση έγινε σήμερα και αύριο πρέπει να ψηφίσουμε. Αν μετά τη σημερινή συζήτηση υπάρξει κάποια πολύ μεγάλη ανάγκη για περαιτέρω τροπολογίες, θα πρέπει να γίνουν προφορικές. Δουλέψτε με τις πολιτικές ομάδες ε, ανάλογα αν θέλετε να υποβάλλετε προφορική τροπολογία, να το πάτε μέσω της πολιτικής ομάδας, να μην έχουμε προβλήματα αύριο. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε την ε, έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ και για τη συζήτηση και για την παρουσίαση. Λοιπόν, έχουμε τώρα χρόνο και για την επόμενη, για την οικοκαινοτομία, το ΓΕΝΣ και οι σκιώδεις να είναι σύντομοι. Και θα έχουμε κατάλογο ομιλητών, αλλά σκεφτείτε αν θέλετε να μιλήσετε. Θέλω να περιορίσω το χρόνο των ομιλητών για να προλάβουμε. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ρωτάει ο μιλητής αν μπορεί να μιλήσει σου ειδικά. Γίνεται. Λοιπόν, αυτή η γνωμοδότηση που ζήτησε η ΕΝΒΗ σημαίνει ότι με την περιβαλλοντική πολιτική μπορεί κανείς να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Και όλοι έχουμε πολύ φιλόδοξες ατζέντε για το περιβάλλον. Πρόκειται κυρίως να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να το διασώσουμε, γιατί τον πλανήτη πρέπει να τον μπορέσουμε να τον παραδώσουμε σε σχετικά καλή κατάσταση σε επόμενες γενναίες. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της ατζέντα του θεματολογίου του φιλόδοξου. Και στην Ευρώπη πρέπει να σκεφτούμε πώς θα λειτουργήσει σωστά η πολιτική για να δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας. Έχουμε μηχανισμούς και μέσα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αρχίσουν αυτές οι διαδικασίες και πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι καινοτόμοι περιφέρειες να ασχοληθούν με όλα αυτά. Οι οικοκαινοτομίες μας βοηθούν, για παράδειγμα, να περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων. Μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματικότερη έτσι τη χρήση των πρώτων υλών. Και όλα αυτά δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Το ξέρω εκ και από τα ορυχεία της Βόρειας Σουηδίας αλλά και από τη δασοκομεία και από τον κλάδο του τουρισμού ε, υπάρχουν συνεχιζόμενες εργασίες με σκοπό α, βιώσιμης παραγωγής. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, η IKEA είναι ένα παράδειγμα, εκεί λειτουργούν με περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία απαιτούν από τους προμηθευτές τους δεν μπορούν όλοι να ανταποκριθούν, αλλά όποιος θέλει να δημιουργήσει νέες δυνατότητες παραγωγής ε, θα αναλάβει μια ε, δουλειά. Οι στατιστικές δείχνουν ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας, αλλά ότι η δυναμική είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε δει μέχρι τώρα. Οι οικοκενοτομίε λοιπόν θα πρέπει να υποστηριχθούν ακόμη περισσότερο μέσα από τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτουμε. Και αυτό συνάδει και με την πολιτική συνοχή, με το, την πολιτική για το 2020 και όλα αυτά ευθυγραμμίζονται και με αυτά που λέγαμε παλιότερα στην Επιτροπή μας σχετικά με το προγραμματισμό της επομένης περίοδου. Οι περιφέρειες πρέπει να ε, υιοθετήσουν στη στρατηγική τους και οικοκαινοτομίες και αυτό ισχύει και για τη λεγόμενη έξυπνη εξειδίκευση, smart specialization. Οι περιφέρειες μπορεί να κάνουν εδώ πολύ περισσότερα πράγματα και πρέπει να υποστηριχθούν. Και αυτό πρέπει να το πούμε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό προσπαθώ να το κάνω στην γνωμοδότηση. Και είμαι και ευγνώμων για τις θεατροπολογίες που μπορεί να βελτιώσουν αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ Γένς ένα σχόλιο και ο Γιάνν Όλμπρεχτ μπορεί να το επιβεβαιώσει. Χθε καταφέραμε να πείσουμε το Συμβούλιο να στηρίξει τις οικοκαινοτομίες ε, του ΕΚΠΑ. Τέσσερις μήνες μάχης χρειάστηκε για να πιστούν για αυτό το πράγμα. Βλέπω ότι δεν είναι εδώ οι αλλά υπάρχουν ε, συνάδελφοι που τους αντικαθιστούν. Για τον Τόμας Ντόιτς από το ΕΛΚ ποιος θα μιλήσει. Κανείς. Εντάξει, πάμε στον, στην Άλντε για τη Φορήκα. Ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Πολύ λίγα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νίλσον για τη δουλειά αυτή. Η κυρία Πακορίνεν τα λέει αυτά. Ευχαριστή. Δεύτερον, η κυρία Πακορίνεν θέλει να υπογραμμίσει το θέμα των ανεκμετάλλευτων ε, δυνατοτήτων που έχουμε για την καινοτομία, την οικοκαινοτομία, που είναι ένα ε, στοιχείο ενεργητικού για την ε, Ευρώπη, για τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης ότι οι νέες καινοτομίες, οικοκαινοτομίες συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη και διατηρήσιμες θέσεις εργασίας. Πολλά θετικά ε, έχει να πει η κυρία Πακορίνεν και εγώ ε, τα υποστηρίζω. Εκεί ε, κατάλαβα από την έκθεση ότι ακόμα είμαστε στον παλιό κανονισμό που θέτει προτεραιότητες και εξετάζει τον αντίκτυπο σε οικολογικό επίπεδο. Ίσως ε, μπορούμε ε, σε αυτό το σημείο να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να δούμε πώς η νέα νομοθεσία θα υποστηρίξει την κατεύθυνση αυτή ε, γιατί όπως είπε και η Πρόεδρος έγιναν πρόσφατα αλλαγές μετά από τη μάχη που δόθηκε στον τριμερή διάλογο. Και τέλος η Σκιώδης λέει ότι πρέπει να έχουμε ε, συγκεκριμένες δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια και την συμφόρηση αν θέλετε που παρουσιάζεται στην εμπορευματοποίηση της οικοκαινοτομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ εμείς ευχαριστούμε. Ανιούς Χρυσόγελος για τους πράσινους. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρος. Ε, η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε καινούριε προσεγγίσεις και στα θέματα της οικονομίας και της απασχόλησης. Και η ε, καινοτομία, δηλαδή η οικολογική καινοτομία, προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και για ανάπτυξη νέων μορφών οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και για ανάπτυξη θέσεων εργασίας, για δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο κύριος Μπαρόζος στην Ολομέλεια πριν περίπου ένα χρόνο είχε πει ότι 20 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας και άρα σε τομείς που έχουν οικολογική καινοτομία σε σημαντικό βαθμό. Αλλά χρειάζεται η οικολογική καινοτομία να ενσωματωθεί στην περιφερειακή στρατηγική και στην πολιτική συνοχή. Δηλαδή, αν δεν μπει στην ε, αντίληψη και των περιφερειακών αρχών και στο σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο, αλλά παραμένει ένα ξεχωριστό αντικείμενο, τότε χάνουμε πολλέ ευκαιρίε και δυνατότητε που έχουμε για να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Σα αναφέρω μερικά παραδείγματα στον τομέα των ορυκτελέων στη χώρα μου. Υπάρχει πολύ αναπτυγμένη τεχνολογία που παίρνει τα παλιά ορυκτέλεα από τα οχήματα και φτιάχνει νέα ορυκτέλεα που είναι υψηλών προδιαγραφών και δεν έχουμε απώλεια πρώτων υλών και έχουμε μείωση της ρήπανσης. Να μια οικολογική καινοτομία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Στον τομέα του νερού σπαταλάμε πάρα πολλά χρήματα για να πάρουμε νερό στις πόλεις από πολύ μακριά. Αλλά θέλουμε οικολογικές λύσεις για μέσα στις πόλεις, για επαναχρησιμοποίηση του νερού, για ανάκτηση του νερού ε, που έχει χρησιμοποιηθεί κλπ. Στο θέμα της ενέργειας δεν έχουν όλες τις περιοχές πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, όμως εκεί υπάρχει τεράστιος τομέας και όχι μόνο με αυτά που βλέπουμε σήμερα να εφαρμόζεται, για παράδειγμα ανεμογεννήτρες ή φωτοβολταϊκά, υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα σήμερα τα οποία πρέπει να γίνουν πράξη που αξιοποιούν για παράδειγμα φυσικές χρωστικές που υπάρχουν στα φυτά για να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Σκεφτείτε μια καινοτομία που θα βάφουμε το σπίτι ή το όχημα και με ειδικά χρώματα τα οποία θα μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας τεράστιος τομέας γι' αυτό που λέμε ότι θέλουμε μια έξυπνη και περιεκτική και ε, βιώσιμη ε, ανάπτυξη αλλά πρέπει να συνδέσουμε αυτά τα θέματα ε, και όπως είπε και η Πρόεδρος χρειάστηκαν μήνες διαβουλεύσεων για να γίνει αντιληπτό και εγώ πολλέ φορέ επέμενα όταν στάγαμε τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχή να προσπαθώ να ε, ενσωματωθούν αυτέ οι αρχέ γιατί γίνεται πολλέ φορέ μεγάλη σύγχυση μεταξύ μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προστασία των οικοστημάτων με την έννοια οικολογική καινοτομία. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι, η οικολογική καινοτομία σημαίνει μια καινούργια δυναμική. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να περιορίσουμε τι περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I am actually shocked, Jens, but nobody wants. Σοκάρομαι, Jens, ε, ε, I would like to give you the floor if you want to... Οπότε ε, δεν ζητεί κανείς το λόγο, πάρε εσύ το λόγο για να κλείσεις το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και θα είμαι ευγνώμων και περιμένω και τις προτάσεις σας μέσα από τις τροπολογίες. Για τις τροπολογίες πρέπει να αποφασίσουμε πολύ γρήγορα δυστυχώς την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών γιατί η διάσκεψη των Προέδρων στο Κοινοβούλιο πήρα απόφαση οι συνεχιζόμενες διαδικασίες ε, για εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας ήδη, που ήδη έγιναν και που ξεπερνούν το εξάμεινο θα ολοκληρωθούν και οι εκθέσεις πρέπει να τελειώσουν μέχρι την 1η Ιουνίου φέτος. Οπότε όλες οι επιτροπές επιτάχυναν πάρα πολύ όλες τις εκθέσεις και το ίδιο πρέπει να γίνει και με τη δική μας τη γνωμοδότηση. Δυστυχώς η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων όταν ε, θα δώσουν ε, από την ΕΝΒΗ θα ληφθεί 6 Ιουνίου και δεν μπορούμε να περιμένουμε γιατί θα ψηφίσει αμέσως η ΕΝΒΗ στον Ιούνιο και δεν θα μπορεί να αναβάλει για την προετοιμασία της δικής μας νομοδότησης. Οπότε 30 Μαΐου είναι η 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία κατάθεσης. Οπότε προσαρμοστείτε ανάλογα 6 το απόγευμα αύριο και θα πρέπει έγκαιρα να δώσουμε την γνωμοδότηση ε, αφού αποφασίστηκε αυτό από τη διάσκεψη των Προέδρων. Και με αυτά κλείνω το σημείο και προχωρώ. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, ο Χόρκια είναι εδώ. Ε, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 6 νωρίτερα. Πάμε στο σημείο 6 λοιπόν. Συνέπειες των δημοσιονομικών περιορισμών για τι τοπικές αρχές όσον αφορά τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης στα κράτη-μέλη. Η κυρία Ερμίνα Ματζόνη κάλεσε δύο εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν και εκείνη τι απόψεις. Φαντάζομαι θα ακούσουμε πρώτα τους εμπειρογνώμονες και μετά θα παρουσιάσετε την έκθεση. Δύο εμπειρογνώμονες έχουμε, τον κύριο Χόρχε Νούνες Φερέρ, ο οποίος είναι συνεργάτης ερευνητής του ΣΕΠΣ, που είναι το Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας της Ένωσης, και τον κύριο Μάριο Μουστήλη, καθηγητής Οικονομικών και διοίκησης από το δεύτερο Πανεπιστήμιο της Νάπολης. Ο Χόρχε έχει πρώτο το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Έρθω να σας μιλήσω. Έχω ασχοληθεί αρκετό καιρό με τα κινητικά ταμεία και τώρα είμαι συντονιστής για την πλατφόρμα SEPS και ξέρω επομένως τα περισσότερα Να σας πω ε, τα εξή. Έχω διαβάσει το έγγραφο εργασία, αυτό το οποίο αφορά την περιοδική πολιτική και τη συνοχή. Είδα τι μηνύματα έχετε εκεί, έτσι προτίμασα την προσφυγή μου. Για να δούμε. Ξεκινώ. Το μήνυμα είναι ότι έχουν παροξυνθεί οι αδυναμίες που υπήρχαν. Βλέπετε εδώ σε αυτό το γράφημα ότι οι περιφέρειες που ταχύτερα ανεπτύσσονται πριν την κρίση είναι αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο, που έχει συρρικνωθεί περισσότερο το ΑΕΠ με την κρίση. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί όταν ο κόσμος ε, μιλάει την κρίση λέει πω όλα τώρα είναι πιο δύσκολα αλλά το θέμα είναι ότι μερικές ε, αυτές τις χώρες, αυτές τις χώρες αυτές τις περιφέρειες ε, τώρα είναι σε χειροτερή κατάσταση, επομένως κάτι θα πρέπει να, να σκεφτούμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε κάποια ζητήματα για τα οποία έχουμε κάποιες ε, κεφαλαιοκές ροές, έχουμε αυτές τις ροές, τις εισροές, έχουμε κάποιες επενδύσεις, έχουμε κάποια δάνεια. Αυτά όμως δεν είναι παραγωγικές ε, κινήσεις. Δεν αφορούν τους παραγωγικούς τομείς. Επομένως, αυτό που το, οποίο είναι πάρα πολύ ε, φανερό, έντονο, είναι το πόσο έχουμε αυτόν τον αρνητικό πληθωρισμό στις τιμές της στέγης στη Γερμανία τα τελευταία 30 χρόνια. Όμως αυτό είναι η, μια στρεβλή ανάπτυξη. Ας είμαστε επομένω πάρα πολύ προσεκτικοί με το πώς το πραγματίσουμε την πολιτική μας. Οι στρατηγικές ακόμα βασίζονται στις υποδομές. Θεωρείται ότι έτσι θα έχουμε ανάπτυξη και όσον αφορά την πολιτική συνοχής αλλά έχουμε πάρα πολύ μείνει πίσω όσον αφορά σε αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε κάνει. Γιατί η στατική της Λισαβόνας δεν εφαρμόστηκε με τρόπο δυναμικό. Θυμάμαι τι, πώς είχε προειδοποιήσει η Κομισιόν την Ιρλανδία, ότι αν κάτι πάει στραβά, τότε η χώρα είναι πολύ εκτεθειμένη. Όχι, έλεγε η Ιρλανδία, όλα πάνε μια χαρά, μην αναμειγνύεστε στα εσωτερικά μας. Αυτά έλεγε η Ιρλανδία τότε στην Ισπανία. Όμως, είδατε τι έγινε λίγα χρόνια αργότερα. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά με το σύμφωνο για την ανάπτυξη. Όμως θα πρέπει πρώτα πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για έξοδο από την κρίση. δεν θα είναι εύκολη η έξοδος από την κρίση. Είναι σημαντικό να επιφέρουμε συστημικές μεταβολές. Ο κόσμος λέει ότι θα πρέπει αυτές οι αλλαγές να επιβληθούν στις περιφερειακές αρχές. Επίσης, όσον αφορά τη μόχλευση του ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση. Και αυτό σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρξουν πόροι. Αλλά να μην ξεχνάτε ότι η μόγλευση γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι δοθεί θα πρέπει να επιστραφεί. Και βέβαια τι κάνει το δημόσιο, μετακυλεί όλα αυτά τα έξοδα που πρέπει να καταβάλει τελικά στον καταναλωτή, στον πολίτη. Όμως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους φόρους. Χρησιμοποιούνται οι φόροι για να καλυφθεί το έλλειμμα, οπότε έχουμε ταυτόχρονα και ψηλότερα τέλη και ψηλότερους φόρους. Αυτό δεν προϊονίζει καλά πράγματα για το μέλλον. Δηλαδή, δεν πάμε να γίνουμε μόνο Αμερικανοί, πάμε να γίνουμε ταυτόχρονα και Αμερικανοί και Δανείοι όσον αφορά την οικονομική μας ε, πολιτική. Ή το ένα όμως ή το άλλο πρέπει να γίνει. Οπότε, έχουμε όλα αυτά τα, τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνοι. Ε, κάθομαι και ακούω τι συζητάτε εδώ, τι αποφάσεις λαμβάνονται ή δεν λαμβάνονται για τον προϋπολογισμό. Οι περιφέρειες, άλλες πιο δραστήριες, άλλες λιγότερες. Θα πρέπει πάντως να αναλάβουν πρωτοβουλίες και σε τοπικό επίπεδο. Δεν θα πρέπει την τελευταία στιγμή και στο γόνατο να ετοιμάζουμε κάποια προγράμματα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μηχανισμός. Ε, εντάξει, να υπάρχει κάποια χρονική στέρηση. Αλλά εάν δεν το φροντίσουμε αυτό, τα προγράμματα θα είναι απονευρωμένα. Και αυτό δεν μας βοηθάει. Και δεν βοηθάει σε τόσο κρίσιμη στιγμή. Πολύ ωραία να μιλάμε για την ενέργεια και για το κλίμα, αλλά καινοτομία, παιδεία, επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν. Θα πρέπει να γίνουν πιο ανθεκτικές οι οικονομίες μας. Είναι αυτό το πρόβλημα με το παρελθόν ακόμα και με την πολιτική συνοχή είναι. Α, λέει ο κόσμος ότι χρειάζεται μια πολιτική συνοχής, διαρκής. Και δεν είναι θέμα μόνο χρημάτων, είναι θέμα στρατηγικής. Να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος στο μέλλον να μπορέσουμε να κάνουμε τις οικονομίες μας πιο θωρακισμένες. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ούτε την Ισπανία ούτε την Ελλάδα. Ακολούθησαν κάποια μοντέλα τα οποία ίσχυαν τότε, τώρα όμως δεν ισχύουν. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερη ευελιξία, να έχουμε και καινοτόμα εργαλεία χρειάζεται να είμαστε και πιο, πιο θαραλέοι, πιο τολμηροί στις επιλογές μας. Πέραν των όσων λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα σημειώματά της, στα έγγραφα εργασίας. Έχουμε αυτά τα ομόλογα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και από πόλεις. Δεν είναι δημοτικά τα ομόλογα αυτά. Είναι κάποια ομόλογα τα οποία συνδέονται με έργο, ομόλογα έργων. Έτσι το έργο είναι εγγυητής για το ομόλογο και εγγυητής για το έργο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται ισχυρά δυναμικά εργαλεία. Υπάρχουν τομεί στους οποίου μπορούμε να... Α, αυτό τώρα πρέπει να επιταχύνουμε όμως γιατί δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το χρονικό όριο. Τώρα κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Είναι ότι ο ιδιωτικό τομέα που έχει εμπλακεί, αυτό είναι κάτι το θετικό, είναι σημαντικό. Χρειάζεται κατανομή εργασίας για να δούμε ποιος και τι θα χρηματοδοτήσει. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Χρειάζεται προσαρμογή, είπαμε. Έχουμε τώρα την μετακύληση, είπαμε, του, του, του, του κόστου αυτού του καταναλωτή. Υπάρχει αυτή η μεσονομική πίεση. Γιατί έχουμε τον ένα φόρο μετά τον άλλο που επιβάλλονται. Πασχίζει κάθε χώρα να βρει τα χρήματα που χρειάζονται από τον καταναλωτή, από τους ίδιους με τους φόρους. Άρα χρειάζεται να προβληματιστούμε σε βάθος. Δεν είναι ο τομέας μου η φορολογία, αλλά σας ξαναλέω ότι αυτή η μέθοδος είναι ανησυχητική πολύ. Θα δούμε επόμενος πώς οι δημόσιες προμήθειες και διαγωνισμοί θα αναθεωρηθούν εκ βάθρων. Πώς το κόστος και το όφελος θα ληφθούν σωστά υπόψη. Πώς επίσης θα αναθεωρηθεί εκ βάθρων το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων. Να ρίξουμε ματιά στο τι γίνεται με τους ανταγωνιστές μας. Να σταματήσουν να μεταξύ μας επίσης. Κάτι να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε επομένω τον ανταγωνισμό των έξοδων. Ας γίνουμε ισχυρότεροι. Ας μην έχουμε μόνο την κόντρα Γερμανίας-Γαλλίας. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με τον έξω κόσμο. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο καθηγητής Μάριο Μουστήλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Έχω ασχοληθεί με την εφαρμογή ευρωπαϊκών ε, προγραμμάτων όσον αφορά την ε, συγχρηματοδότηση ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε τα ευρωπαϊκά ταμεία που μπαίνουν στη λογική της συγχρηματοδότησης στα πλαίσια του 1320, 2013-2020. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διχοτόμηση των ε, δημοσιονομικών πολιτικών που σχετίζονται με το δίκτυο ανάπτυξης και ένα πιο τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με τον τρόπο που ε, αυτό τα σχέδια μπορούν να μας δώσουν μία συνοχή με τις οικονομικές ε, πολιτικές. Και έτσι μπορούμε να έχουμε να κάνουμε με ένα συμβιβασμό για να μην υπάρχει αυτή η διχοτόμηση των δύο στόχων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποκαταστήσουμε την δημοσιονομική ασφάλεια μέσα στα πλαίσια της ε, αντιμετώπισης των ε, ομολογιακών δανείων που έχουμε αναλάβει. Το θέμα δεν αφορά την αλλαγή στρατηγικής ή κατεύθυνσης, αλλά την χρονική εφαρμογή των προγραμμάτων, δηλαδή την επιτάχυνση ε, απόδοσης χρέους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την στρατηγική σε όλες τις χώρες. Οι πρόσφατες αναλύσεις σχετίζονται με αυτό τον πυλώνα στον οποίο βασίζεται η λιτότητα, η λιτότητα των δημοσίων οικονομικών. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην είμαστε ε, self-defeating, δηλαδή να μην είμαστε ητοπαθείς ε, αφεαυτοί. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την δημοσιονομική συρρήκνωση έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης του χρέους. Αυτό έχει να κάνει και με τον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση του output οδηγεί στο κεινσιανικό πρότυπο της παγίδας της ρευστότητας. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει καμία χρηματοδότηση. Τα asset δημιουργούν καταβαράθρωση και το λεγόμενο credit crunch, μειώνεται η ζήτηση ε, και φτάνουμε σε μια πιστοτική ασφυξία, credit crunch. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε σε αυτά τα πλαίσια και, τα ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Ίσως λοιπόν αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να δούμε κατά πόσο σταθεροποιήθηκαν τα spread, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι ισχύει και για την Ιταλία. Η συρρήκνωση της οικονομίας περνά από την συρρήκνωση των εισαγωγών. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε ισοσκέληση των προϋπολογισμών σε σχέση με το δημόσιο χρέος. Αλλά τι θα κάνουμε ως προς την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Η οικονομία πλήθεται άρδιν και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η βιώσιμη ανάπτυξη χωρών όπως ε, η Ιταλία και η Ισπανία. Έχουμε μία μείωση του παραγωγικού δυναμικού που μπορεί να φτάσει ε, πολύ υψηλά ποσοστά. Μέσω πρόθεσμα λοιπόν έχουμε να κάνουμε μία συρρήκνωση της Ιταλικής οικονομίας, κάτι το οποίο θα αποδυναμώσει και παραγωγικούς τομείς όπως και τις εξαγωγές. Υπό το φως αυτών των σκέψεων προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε επιλεκτικές πολιτικές αντιμετώπισης των δαπανών Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα ορίσουμε το output μας ε, μέσα στα πλαίσια μίας εξυγίανσης. Η νομισματική πολιτική είναι ε, αρκετά επεκτατικής μορφής και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο η νομισματική πολιτική μπόρεσε να αντιμετωπίσει και θέματα αποπληθωρισμού. Γι' αυτό, ε, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις προσταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι η λιτότητα πλήττει περισσότερο τις χώρες στην οποία εφαρμόζεται μηχανικά ή μηχανιστικά. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτό το φαύλο κύκλο της εξυγίανσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ε, μία δημοσιονομική εξισορρόπηση. Τα οικονομετρικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σήμερα ακόμα και από την ε, Κομισιόν χρησιμοποιούν δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές μέσα στα πλαίσια της αντιμετώπισης της οικονομικής ε, κρίσης της τάξης του 0,5%. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τη ζήτηση. Όμως το, ε, διεθνώς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είδε ότι οι πολλαπλασιαστές σήμερα είναι της τάξης του 0,5% από 0,5 έως 1,7. Άρα έχουμε μία συρρήκνωση της οικονομίας η οποία διπλασιάζεται. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λαμβάνει υπόψη ε, μέτρα τα οποία είναι αντιπαραγωγικά. Γι' αυτό θα πρέπει να τεθεί εκ νέου η συζήτηση μέσα στα πλαίσια ενός ε, δημοσιονομικού συμβολέου. Ποια είναι η βάση του Fiscal Compact. Εάν αυξηθεί το δημόσιο χρέας, τότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ελέγξουμε τις δαπάνες, διότι μειώνεται η κατανάλωση. Εάν όμως το δημόσιο χρέος δεν αυξηθεί, τότε θα κατεβληθούν και λιγότεροι φόροι για τον έλεγχό του. Είναι πράγματι έτσι μπορούν να υπάρξει νέα εμπιστοσύνη στις αγορές με βάση αυτή την φορολόγηση και την ε, δημοσιονομική πολιτική. Νομίζουμε ότι δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Μπορούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του δημόσιου χρέους κατά αυτό το τρόπο. Ακόμα και εάν υπάρξει αυτή η συνεχής ανάπτυξη θα μπορούσαμε να έχουμε ανάπτυξη του ΑΕΠ υψηλότερη από αυτή του χρέους. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα μπορούσε να επιληθεί με διαρθρωτικές αλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη που να μην σχετίζονται με το Fiscal Compact. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα η πρόταση να αποκλείσουμε το, ε, το μοντέλο σταθερότητας και το σύμφωνο σταθερότητας μέσα στα πλαίσια αυτής της στενής δημοσιονομικής αντιμετώπισης της ε, κρίσης. Γι' αυτό και τα σχέδια συνοχής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι συσταλτικά, αλλά διασταλτικά. Και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εναλλεκτικές που μπορούν να εξευρεθούν. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στο τμήμα εκείνο της ε, συγχρηματοδότησης που αφορά τις ε, καθαρές εισρωές και εις πράξεις του κράτους, όπως το ΦΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα σχέδια να γίνουν ε, ε, βιώσιμα έτσι ώστε να υπάρξει και σωστός χρονισμός της ε, χρηματοδότησης από το εθνικό επίπεδο και από το ευρωπαϊκό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σωστός χρονισμός και κατά τα τελευταία έτη του προγράμματος τότε να χρησιμοποιηθούν μόνο τα εθνικά κονδύλια. Στην αρχή να βασιστούμε στη συγχρηματοδότηση για να έχουμε ε, καλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης και ε, υψηλότερου δίκτυ του ΑΕΠ. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε έναν πραγματικό προγραμματισμό των επενδύσεων, όπως καταδεικνύουν και ορισμένοι τομείς. Εάν όμως επιλέξουμε καλύτερα και προγραμματίσουμε καλύτερα τις παρεμβάσεις μας, τότε θα μπορούσαμε να έχουμε μία διαφορετική χρηματοδοτική πολιτική η οποία ε, να ισχύσει πρωτίστως σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναντι των ε, κρατών μελών. Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε. Και τώρα ο συνάλφος Ρόκο Μπουμπίκο από την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, αν θέλετε, σε αυτό το στάδιο να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, η έκθεση είναι καταπληκτική ευκαιρία για μας να παρουσιάσουμε απόψεις για τις γενικές τάσεις που είδαμε και αναλύσαμε τα τελευταία χρόνια πολλές αναλύσεις που κάναμε μέχρι τώρα συμβαδίζει με την ανάλυση της έκθεσης. Στην τελευταία έκθεση για την πολιτική συνοχή θα δούμε την έκβαση όλων αυτών. Επίσης υπάρχουν και κάποια προγράμματα του ΟΣΑ για αποτελεσματικές δημόσιες επενδύσεις από τοπικές αρχές σε δημοσιονομικές, δημοσιονομικά δύσκολες εποχές. Οι προκλήσεις που ακούσαμε αφορούν ε, δύο τομείς που θα περιέχονται στις ανακοινώσεις. Το ένα είναι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και η μακροοικονομική διακυβέρνηση και εκεί θα μιλήσουμε κυρίως για τη σημασία ε, υγιών οικονομικών πλαισίων και πώς ένα υγιές οικονομικό πλαίσιο είναι σημαντικό για τη λειτουργία των ταμείων και το άλλο είναι η σύγκληση προς ε, το μεσοπρόθεσμο στόχο MTO και εκεί πρέπει να δούμε για να αναλύσουμε πώς θα χειριστούμε τη συγχρηματοδότηση στο φως των όσων ακούσαμε επίσης και στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι κινούμεθα μέσα σε όρια. Τα όρια τα θέτει το βασικό σχέδιο για τον μεσοπρόθεσμο στόχο. Αυτό έχει αποφασιστεί από πέρσι. Ε, η ρήτρα της επένδυσης πρέπει να είναι προαιρετική και να υπάρχει στα πλαίσια και να λειτουργεί στα πλαίσια των συμφώνων ε, δημοσιονομικού και της ανάπτυξης και δεν μπορούν να υπάρξουν παρεκκλήσεις από το μεσοπρόθεσμο στόχο. Mid-term objective. MTO. Γενικά πρέπει να πούμε ότι τα διαρθρωτικά ταμεία τη συγκεκριμένη εποχή είναι σημαντικά ε, και για τη μεγέθυνση και για την ανάπτυξη επίσης. Και αν δούμε την εξέλιξη του ΑΕΠ και τι ε, μεγενθύνει το ΑΕΠ, μπορούμε ε, να δούμε ότι παντού μπορούν να συμβάλλουν τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδιαίτερα αν μιλάμε για κεφάλαια, ανθρωπίνο κεφάλαιο, παραγωγικότητα ανθρωπίνου κεφαλαίου. Για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία έχουμε μια κέρια συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων. Παράλληλα με την έκθεση Ματζόνη πρέπει να πω ότι γίνεται και πολλή δουλειά τώρα στην Κομισιόν και θα δούμε τα αποτελέσματα ήδη τις επόμενες εβδομάδες όταν θα, εγκριθεί, θα εγκριθούν οι πρώτες ανακοινώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ματσόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι σημερίζεστε την ανάγκη να συζητήσουμε επί μιας έκθεσης που σχετίζεται με τις δημοσιονομικές προσταγές στα πλαίσια του Δημοσιονομικού Συμφώνου και τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ευχαριστώ την Επιτροπή για το ότι εκτίμησε την εργασία μας και γιατί προσπαθεί να βρει ανοίγματα σε σχέση με την αναθεώρηση Τη της ε, διάθεσης ε, κονδυλίων στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που παρενέβησαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση όταν ε, ορίσαμε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές αυτής της έκθεσης και ελπίζω σε αυτό το προσχέδιο να ενταχθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Πρόκειται για ένα ανοιχτό ε, έγγραφο για ε, περαιτέρω συμμετοχές και συνεισφορά. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους που ενίσχυσαν αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ και τους δύο καθηγητές, Φερέρ και Μουστήλη, οι οποίοι ε, συνεισέφεραν ουσιοδός κατά διαφορετικό τρόπο στα πλαίσια της γενικότερης μας ε, θέσης. Βεβαίως η θέση μας ε, δεν είναι καινούρια. Πρόκειται για ένα από τα βασικά ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει καθώς και τις κυβερνήσεις. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο συνεισφέρει με όλες του τις δυνάμεις για έναν πολιτικό διάλογο ύψης της σημασίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση για να δούμε πώς οι, προστα... οι δημοσιονομικές προσταγές μπορούν να βοηθήσουν και πώς ορίζεται η μείωση της παραγωγικότητας, αυτή η τάση που ε, διαγράφεται για τη μείωση της απασχόλησης, τα κράτη δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν το δημόσιο χρέος, όπως βλέπουμε. Και υπάρχει και διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, όπως ε, ανέφερε και ο καθηγητής Φερέρ αυτό το χάσμα, αυτή η διαφοροποίηση μας οδηγούν σε μεγαλύτερες ανησυχίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα spread διαφέρουν από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η πολιτική ε, συνοχής ε, είναι δύσβατη γιατί δεν πληρούνται οι οικονομικοί και κοινωνικοί όροι προς μία σύγκληση. Ελπίζω να ακούσω και περαιτέρω ε, υποδείξεις και βεβαίως ε, ε, δεν δίνουμε μία ολοκληρωτική λύση, αλλά προσπαθούμε να μιλήσουμε για την αναπτυξιακή ανάγκη και μετά τις πολιτικές κυρώσεων προσπαθούμε να ορίσουμε την, ε, μια νέα διάσταση αναπτυξιακών μέσων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που έχει σημασία είναι στα πλαίσια της πολιτικής σύνοχης να δούμε κατά πόσο υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες επενδύσεων, διότι αυτό είναι κάτι το καθόλου αμεληταίο. Ο καθηγητής μου στείλει τονίζει ότι η δυνατότητα επενδύσεων θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία των τοπικών αρχών και θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν τάχιστα και σκόπιμα για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη των ε, περιφερειών, των περιφερειών μας. Άρα προτείνουμε να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα αναθεώρησης των κανόνων για να ορίσουμε δημοσιονομικά κριτήρια τα οποία να είναι σκόπιμα και να μας επιτρέψουν μία πραγματική συγχρηματοδότηση. Οι δαπάνες για την συγχρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να οδηγήσουν στο να υπερβούμε το πρόβλημα των spread που διαφέρουν από κράτος σε κράτος και να μπορέσουμε δημοσιονομικά να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση αντίφασης από την οποία πρέπει να βγούμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε παρά την λιτότητα και παρά την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, γιατί αξιοποιήσατε τάχιστα αυτή την έκθεση, έτσι ώστε αυτή η έκθεση να αποτελέσει μέσο διαπραγμάτευσης για νέους ε, κανόνες που θα ορίσουμε στις επόμενες δημοσιονομικές πολιτικές. For the socialist, ε, ο κύριος για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω τις προτάσεις του Ευγένη Κυρίλοφ, συναδέλφου, που είναι τώρα στην αντιπροσωπεία, ναι, στην Προεδρία στο Προεδρείο. Γι' αυτό τον αντικαθιστώ. Θέλω να πω ότι και εγώ στηρίζω τις ιδέες του. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Ματσόνη για το σχέδιο έκθεσης που πιάνει τις βασικές δυσκολίες και προκλήσεις για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων ε, σε περιόδους ε, δύσκολες θα προτείνω κάποια πρόσθετα θέματα που αφορούν το ζήτημα αυτό για να συμπεριληφθούν στο σχέδιο έκθεσης και θα τα υποβάλω ως τροπολογίες. Συμφωνώ απόλυτα με την ε, ανησυχία που εκφράζει η έκθεση ότι οι ανισότητες ε, μεταξύ ε, φτωχές και πλούσιες χώρες και οι διαπεριφερειακές διαφορές σε πολλά κράτη-μέλη επιμένουν και αυξάνονται. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται κατάλληλα μέτρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κι άλλα δηλαδή. Όμως υπάρχει τάση σε κάποια κράτη-μέλη να συγκεντροποιούνται τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων και έτσι πάμε από την περιφερειακή στην κεντρική διαχείριση. Ε, για καλύτερες ε, δυνατότητες συγχρηματοδότησης και υλοποίησης. Ακόμα και αν έχει νόημα κάποια τέτοια απόφαση, δεν έχει ε, νόημα αν δεν λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε όλη τη διαδικασία υλοποίηση των έργων. Αυτό σημαίνει δηλαδή μεταξύ άλλων το κεντρικό επίπεδο πρέπει να κάνει πιο πολλέ προσπάθειε για να βρει λύσει για τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των περιφερειών και να εγγυηθεί ισόρροπη κατανομή των ενωσιακών κονδυλίων ε, και για την εθνική συγχρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε ε, να εφαρμοστεί η αρχή της εταιρική σχέσης. Χωρίς αυτή, ε, σε όλα τα επίπεδα τα σημαντικά, υπάρχει μεγάλη, ε, μεγάλος κίνδυνος να επιδεινωθεί η κατάσταση στις περιφέρειες και σε κάποια κράτη-μέλη επίσης. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε στην έκθεση κάποια γνωστά προβλήματα που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη καλύτερης διοικητικής ε, και θεσμικής ικανότητας να, αντιμετωπίζονται τα προγράμματα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και καμιά φορά και σε κεντρικό επίπεδο. Όταν υπάρχουν λιγότερα χρήματα είναι σημαντικό τα διαθέσιμα κονδύλια να δαπανώνται σωστά έγκαιρα και με τρόπο τέτοιο ώστε να πιάνουν τις βασικές προτεραιότητες και ανάγκες. Και εδώ ήρθε η ώρα να σας πω για μια πληροφορία που μας ήρθε χθε το βράδυ μετά από μια εκδήλωση που οργανώθηκε με, το, με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Ινστιτούτο Έργων που δείχνει τα κενά και τις ελλείψεις που έχουμε στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις παγκόσμιες τάσεις και τους παγκόσμιους ανταγωνιστές. Δεύτερον, η διοικητική ικανότητα είναι ο καλύτερος τρόπος για καλύτερη χρήση των υφισταμένων κονδυλίων και πόρων και ε, να αυξήσουμε την ικανότητα των περιφερειακών και τοπικών εμπλεκομένων να συμμετέχουν στα έργα και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα έργα αξιοποιώντας τους ε, λιγοστούς μας πόρους σήμερα. Δεύτερον, η γραφειοκρατία, οι σύνθετοι κανόνες και διαδικασίες, γραφειοκρατία μαζί με οικονομικές δυσκολίες περιορίζουν τη θετική έκβαση της χρήσης των ενωσιακών κονδυλίων. Είδαμε τι σημαντικό ρόλο παίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε δύσκολες περιόδους, πώς στηρίζει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες για να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα χρήματα που τους δίδονται. Μπορούμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή της Τράπεζας Επενδύσεων με πραγματογνωμοσύνη, τεχνογνωσία για να βοηθηθούν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε προτάσεις και αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτά είχα να σας πω ε, για λογαριασμό του Ευγέννη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ε, για τους φιλελευθέρους τώρα. Good Thank you, Chair. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα αλλιώς να είναι τα πράγματα, αλλά δυστυχώς η αλήθεια αυτή είναι πικρή. Θέλει να εξαιρέσει εδώ ο συνεισηγητής την συγχρηματοδότηση από τις παραμέτρους του Συμφώνου Σταθερότητας. Αυτό όμως σήμερα δεν είναι εφικτό και ούτε αύριο θα είναι εφικτό, διότι ανοίξετε μία ματιά ακριβώς στο νομοθέτημα που έχουν 25 χώρε εκτός από Τσεχία και εμένα που υπογράψει εκεί λέει ξεκάθαρα τα εξή αυτό το σύμφωνο ότι θα πρέπει όχι στο 3, 0,5 του ΑΕΠ θα πρέπει να φτάσουμε και μιλούμε για τρεις μονάδες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εάν το έλλειμμα είναι υψηλότερο, μεγαλύτερο. Και αυτό το οποίο κανεί θα μπορούσε να επικαλεστεί τώρα είναι η απόφαση του Συμβουλίου του 2005. Ο κανονισμός 1056. Εκεί δηλαδή, σε εκείνους τους τομείς της οικονομίας που έχουμε την επιβράδυνση. Δεν είναι δυνατόν επομένω η συγχρηματοδότηση να εξαιρεθεί από τις παραμέτρους του Συμφώνου Σταθερότητας. Επομένω, αυτό που θα πρέπει κανείς να τονίσει στην έκθεση και να αναδείξει είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει το σύμφωνο. Όμως δυστυχώς το σύμφωνο έχει κυρωθεί, εγκριθεί πάρα πολύ πρόσφατα αυτές τις, όλες αυτές τις επομένω. χώρες Θα πρέπει να λάβει υπόψη το ότι εκτός από την επιβράδυνση θα πρέπει να ληφθεί και υπόψη το ότι χρειάζεται συγχρηματοδότηση. Και αν κανείς συγχρηματοδοτεί, τότε θα πάει το έλλειμμα πάνω το 0,5%. Οτιδήποτε άλλο πούμε σημαίνει ότι ζούμε σε, σε άλλο πλανήτη. Δηλαδή, άλλα θα πει η Οικονομική Επιτροπή, άλλα εμείς. Ε, τελικά όλα αυτά είναι ευσεβείς πόθη, αν τα πούμε. Επίσης, για αυτή την μακροοικονομική αιρεσιμότητα που είναι το σημείο παριθμών 12 εδώ έχω να σας πω κάτι στο οποίο είναι κατά ο εισηγητής ενώ γνωρίζει τι πρεσβεύει το Συμβούλιο και τι πρεσβεύει και η Κομισιόν η μακροοικονομική εξάρτηση μπορώ να σας δώσω στοιχεία τα οποία κατατείνουν ότι από το 2009 μέχρι το 2013 δεν υπάρχει κανείς συσχετισμός της ποιότητας της απορρόφησης σε σχέση με το έλλειμμα. Οπότε, θεωρητικά, καλά τα λέει κομισιόν, αλλά είναι ατεκμηρίωτα όλα αυτά. Αυτά κανείς θα μπορούσε να προσθέσει στην έκθεση και έτσι να είναι ακριβέστερα όσα προτείνονται. Τρίτον, αυτό το οποίο θέλω να προτείνω στην, στην εισηγητρία είναι το ότι σε αυτήν την έκθεση δεν υπάρχουν στοιχεία για την προσθετικότητα. που είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ σοβαρό για κρατημέλη και περιφέρειες ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να αποκριθεί σε αυτό το οποίο ζητείτε εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που λέει ότι για την περίοδο 2010-2013 έχουμε την προσθετικότητα, δηλαδή ποιο είναι το επίπεδο της αναφοράς πέραν της χρηματοδότησης. Όλες οι χώρες θα πρέπει να μπορέσουν να προβούν σε χρηματοδότηση επενδύσεων. Μιλάμε για 94 δις. Αυτό είναι το επίπεδο αναφοράς. 22-23% αν υπολογίσετε. Θα δείτε πόσο αυτές οι επενδύσεις ωφελούν σε εθνικό, σε τοπικό επίπεδο, θα καταλάβετε ωφελούν αυτές οι επιπλέον πληρωμές. Πάντως θα πρέπει να λάβει υπόψη η συγκέντρια για το ότι θα πρέπει μέσω πρόθεσμα να δούμε τι αποτελέσματα έχουμε και θα πρέπει να κάνουμε αυτή την επαλήθευση το 2012 και εκεί μπορείτε να διπιστώσετε τα εξή ενδιαφέροντα ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες πάρα πολύ μείωσαν την δημόσια χρηματοδότηση, δημόσιες δαπάνες, 20, μέχρι 22, 21, 23%. Τέσσερις χώρες βλέπω εδώ τουλάχιστον και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αύξησαν τις δαπάνες. 52% η Ισπανία. Η Ιταλία Η Πολωνία 57%, Σλοβακία 59%. Άρα κάποιες χώρες αυξάνουν το κομμάτι της ανεξάρτητης επιπλέον επένδυσης και σε περιφερειακό Σε κάποιες χώρες όμως το αντίθετο. Η Επιτροπή συμφώνησε λόγω κρίσης. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο το ότι το πρόβλημα αυτό δεν το έχουμε θίξει ποτέ στην Επιτροπή μας. Και ίσως και γι' αυτό και εσείς δεν είπατε τίποτα στην έκθεσή σας. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο πρέπει να το αναλύσουμε. Πώς πέραν της συγχρηματοδότησης έχουμε την επιπλέον χρηματοδότηση την οποία εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδάλλως, κανείς δεν έχει όλα τα δεδομένα ούτως ώστε να είναι εντάξει. Όπως λέτε και στην εκθεσή σας. Πρόκειται για άμεση σχέση και επίπτωση με την κατάσταση όπως διεπιτόρα... Ε, την Ευρώπη σε τοπικό επίπεδο. Εγώ σε ευχαριστούμε μας ότι υπάρχει πρόβλημα τώρα με το διορθωτικό έλλειμμα, αλλά δεν έχουμε όμως τώρα κάποια πιστική θεωρία, κάποια, για ένα πιστικό ορισμό, κάποια μεθοδολογία για να το, για να το υπολογίσουμε εκτός μικροφώνου, Ήβο. Ε, ε, Και τώρα θα δώσουμε τις σκητάλη στον Νίκο Χρυσόγελ για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που στάμε τώρα γιατί άπτεται τη δυνατότητας των οικονομιών και ιδιαίτερα των, περιφερειών να βγούμε από την κρίση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα, ότι έχουμε μία κρίση, η, η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ένταση της λιτότητας και διαπιστώνουμε τώρα όλοι ότι χρειάζονται επενδύσεις για να βγούμε από αυτή την κρίση αλλά την ίδια στιγμή τώρα δεν υπάρχουν οι για να γίνουν επενδύσεις με βιώσιμο τρόπο. Γιατί στην Ευρώπη δεν θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις ε, που είναι βρώμικες, που είναι αυτές που είναι, θα λέγαμε, ε, δεν είναι βιώσιμες κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό που λέμε συνέχεια, έξυπνη, περιεκτική, βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν σε μεγάλο βαθμό περιορίζεται με τις σημερινές πολιτικές. Κοιτάξτε, Παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε ύφεση 25%. Μεγάλη δυσκολία να γίνει η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μειώνεται και σε απόλυτους αριθμούς αλλά και αναλογικά. Πώς μπορούμε λοιπόν να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Δεν υπάρχει τρόπος να βγεις με μεγαλύτερη ύφεση, με μείωση των δαπανών από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και όλα τα χρήματα που υπάρχουν στο πρόγραμμα να πηγαίνουν μόνο για τη χρηματοδότηση και πάλι να μην επαρκούν εμείς για να βγούμε από την κρίση θα έπρεπε να επενδύσουμε στην καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, σε νέους τομείς οικονομίας, σε αποτελεσματική χρήση των πόρων και αυτό χρειάζεται επενδύσεις. Αυτό είναι σίγουρα, αυτό είναι ο δρόμος. Τώρα, θέλουμε νέα εργαλεία. Θέλουμε καταρχήν να αλλάξουμε και πολιτικές, γιατί εάν συνεχίσουμε αυτή την πολιτική δεν βγαίνουμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Ένα απλό παράδειγμα εάν είχε μειωθεί η ύφεση στην Ελλάδα και υπήρχαν βιώσιμες επενδύσεις θα μειώναμε το χρέος 20%. Άρα αν πήγαιναν χρήματα στις επενδύσεις θα πετυχαίναμε δημοσιονομικούς στόχους πέρα από την, βέβαια, την οικονομική αναζωγόνηση και την απασχόληση. Αλλά πού θα βρεθούν αυτοί οι πόροι. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ο ρόλος του δημόσιου τομέα δεν μπορεί να είναι μοναδικός αλλά ο δημόσιος τομέας πέρα από τις επενδύσεις έχει και ένα τομέα ο οποίος λέγεται προμήθεια, συμβάσεις. Αυτός ο τομέας είναι σημαντικός εάν το συνδέσουμε με καινοτομία γιατί μπορεί να δώσει όθηση, αποτελεί μεγάλο ποστό των, ε, της κατανάλωσης 16 με 17% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο τομέας, ο δημόσιος, θα έπρεπε να είναι εργαλείο καινοτομίας οι περικοπές όμως προπολογισμού των περιφερειών και των δήμων και του δημοσίου γενικά από τη μια αλλά ειδικά η στόχευσή τους σε πιο φτηνά προϊόντα και υπηρεσίες αφενός ενισχύει παλιές δομές, παλιές υπηρεσίες λιγότερο αποτελεσματικές, λιγότερο υπεύθυνε περιβαλλοντικά και απ' την άλλη μειώνει τη δυνατότητα καινοτομία. Επίσης ένα σημαντικό θέμα είναι ότι η μείωση του προϋπολογισμού σε περιφέρειες που έχουν μεγάλη εξάρτηση από το κεντρικό κράτος είναι πολλαπλή. Έχουμε στην Ευρώπη διαφορετικές ταχύτητες. Υπάρχουν περιφέρειες που είναι καλά οργανωμένες και αναφέρθηκαν και στην έκθεση ότι αυτές οι περιφέρειες υποκατέστησαν την απώλεια επενδύσεων από, την από το κεντρικό κράτος και εξορόψαν λίγο την κατάσταση. Δηλαδή εκεί που χάθηκαν επενδύσεις από ένα κεντρικό κράτος ήρθαν ορισμένε περιφέρειες και αύξησαν τι επενδύσεις, άρα εξορρόψαν αυτή την κατάσταση. Το πρόβλημα είναι όμως ότι έχουμε πολλές χώρες, ειδικά στο Νότο και στην Ανατολική Ευρώπη, που οι περιφέρειες δεν έχουν ιδίους πόρου και δεν μπορούν να παίξουν το σημαντικό ρόλο αυτό για εξορρόψη. Άρα μειώνονται και οι δικοί του προπολογισμοί και του κεντρικού κράτου Να σα αναφέρω ένα παράδειγμα ο προϋπολογισμός των περιφερειών στην Ελλάδα από ιδίους πόρους είναι 1, 2, 3% των προγραμμάτων τους, άρα είναι πολύ δύσκολο να κάνουν επενδυτική πολιτική και οι απώλειες από τους κεντρικούς πόρους, από το κράτος δηλαδή προς τις περιφέρειες, έχουν μειωθεί κατά 60%. Άρα μπαίνουμε σε ένα θανατηφόρο κύκλο. Για ποια περιφερειακή ανάπτυξη μπορούμε να κάνουμε. Και ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Χάνουν ανθρώπινο δυναμικό είτε γιατί βγαίνει στη σύνταξη είτε γιατί στις συνθήκες εργασίας που υπάρχουν σήμερα το προσωπικό αυτό επιλέγει να φύγει. Άρα τα πιο δυναμικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό εν ώψη της περίοδου 14-20 ή δεν υπάρχουν ή αν υπήρχαν φεύγουν και καταλείπουν τη διοίκηση. Άρα για πώς θα σχεδιάσουμε περιφερειακή ανάπτυξη. Πρέπει να τα δούμε αυτά σε βάθος. Γιατί δυστυχώς λέμε να περάσουμε σε μια νέα φάση επενδύσεων και ανάπτυξης αλλά ενδιάμεσα έχει καταρρεύσει και το ανθρώπινο δυναμικό και οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η μεταστροφή. Και μάλιστα μέσα στο 2013 για να μπορέσουν οι περιφέρειες να πούνε τα σχέδιά τους, να τα ενσωματώσει το κεντρικό κράτος και να υπογράψει τη Σύμβαση εταιρική Σχέσης με την Κομισιόν για ένα βιώσιμο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης. Και να τονίσω επίσης ότι ε, οι περιφέρειες που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες θα υποστούν και μεγαλύτερε επιπτώσει. Δηλαδή αυξάνει το χάσμα και δεν πετυχαίνουμε στη σύγκληση και την κοινωνική συνοχή που θέλουμε μέσα στι πολιτικέ. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε και από τι εκθέσει που έχουν παρουσιαστεί και στη δικιά μα επιτροπή ότι ήδη ορισμένε περιφέρειε στην περίοδο τη αρχική φάση κρίση μετάπεσαν από κατηγορία σε κατηγορία. Ήταν, στην προηγούμενη έκθεση είχαμε δει ότι 9 περιφέρειε έπεσαν στην κατηγορία των ενδιάμεσων. Είμαι σίγουρο ότι ακόμα περισσότερε έχουν υποστεί αυτή την μεταβολή αυτή την ε, περίοδο. Και επίσης και περιοχές όπως είναι τα νησιά χρειαζόμαστε ειδικά σε αυτή την περίοδο της κρίσης και να αποτυπώνουμε την πραγματικότητα που υπάρχει στις περιφέρειες. Πολλές φορές δείκτες όπως είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Επειδή είμαι από περιφέρεια νησιωτική και είμαι και περιφερειακό σύμβουλο, σα λέω ότι πολλά νησιά λόγω των περικοπών στι κοινωνικέ πολιτικέ και στην υγεία δεν έχουν στοιχειώδη πρόσβαση συστήματα υγείας. Κινδυνεύουν να μην έχουν πρόσβαση στις μεταφορές. Άρα για ποια σύγκληση μιλάμε. Και όμως αυτές οι περιφέρειες σαν ΑΕΠ μπορεί να φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ διαφορετική. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Jan ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω κάτι τους εμπειρογνώμονες ε, και να κάνω και μια πρόταση στην εισηγήτρια για τους ε, εμπειρογνώμονες. Νομίζω ότι είμαστε αντιμέτωποι με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έτσι το πω έτσι ακραία. Αν η πολιτική συνοχή είναι το καλύτερο εργαλείο σε περίοδο κρίσης. Είναι ή δεν είναι. Τι ρόλο παίζει η πολιτική συνοχής εν μέσω κρίση. Και όταν λέω πολιτική συνοχής ε, ε, μιλάω για τη μέθοδο, όχι για τα διαφορετικά ταμεία. Έχουμε την επιμερισμένη διαχείριση ω μέθοδο. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει σοβαρή ευθύνη που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Και το θέμα είναι πώς θα διαμορφώσουμε την πολιτική συνοχή στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τη, όλες τις ευθύνες που αναλαμβάνουν και αρμοδιότητες των κρατών μελών στη δημοσιονομική πολιτική, την εξυγίανση κλπ. Ένα συμπέρασμα που αναφέρει και η συγγήτρια είναι ότι τα κράτη-μέλη αντιδρούν πολύ γρήγορα στα πλαίσια της εξυγίανσης και σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία και μειώνουν την ανεξαρτησία του προϋπολογισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για λόγους εξυγίανσης μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αλλά η συνέπεια είναι μια έντονη ε, συγκεντρωποίηση όλης της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν την πολιτική που βασίζεται στην επιμερισμένη διαχείριση, αλλά μεσούσης της κρίσης η πολιτική αυτή ε, γίνεται πολύ περισσότερο κεντρική γιατί η εξυγίανση σημαίνει ότι τα περιφερειακά και τοπικά ταμεία έχουν μικρότερο περιθώριο ελιγμών και συρρυκνώνεται και η ανεξαρτησία τους. Η Κομισιόν μας παρουσίασε τώρα μια σημαντική έκθεση για ε, ενδιαφέροντα προγράμματα σε πόλεις στην Ευρώπη. Ωραία ανάλυση που δείχνει σαφέστατα ότι η επιτυχία των τοπικών έργων σήμερα εξαρτάται από τη σαφήνεια της εθνικής στρατηγικής. Δεν είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο σημαντικά τα έργα, αλλά πρέπει να υπάρχει στρατηγική καλή σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο. Αναπόφευκτη είναι η συγκεντροποίηση της πολιτικής λοιπόν ή όχι. Και ρωτώ, με οικονομικούς όρους. Το θέμα της διακυβέρνησης είναι σημαντικό για όλη την ανάλυση. Δεν είναι το θέμα αν οι τελικοί ε, αποδέκτες παίρνουν τα χρήματα ή όχι και τα διαθέσουν, αλλά ε, ε, μιλάμε εδώ σε επίπεδο συνολικής δομής. Αν μιλήσουμε για τη συγχρηματοδότηση στο Σύμφωνο Σταθερότητας, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό προϋποτίθεται η Συμφωνία των Ευρωπαϊκών Αρχών, όπως ε, ακούσαμε να λέγεται. Υπάρχουν και στη χώρα μου κάποιες προτάσεις που θα συνδέσουν το έλλειμμα σε τοπικό επίπεδο και τον προϋπολογισμό σε τοπικό επίπεδο και τη συγχρηματοδότηση. Τέλος πάντων, Ρωτώ. Θα αλλάξει η φιλοσοφία της διακυβέρνησής μας. Δηλαδή μπήκαμε στη διαδικασία να αλλάξουμε τρόπο σκέψης για την πολιτική συνοχής και την επιμερισμένη διαχείριση. Γιατί χρειάζονται εδώ στεναρές, στιβαρές πολιτικές, ταχείες πολιτικές, μια αιρεσιμότητα, conditionality, που θα έχει σαφείς στόχους για τη μεγέθυνση. Κάποιος που θέτει τους όρους, ας πούμε, ε, βέβαια έχει και αυξημένη εξουσία. Αυτό το ερώτημα τίθεται τώρα για μας. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές περιμένουν τις απαντήσεις, γιατί η τάση είναι ξεκάθαρα συγκεντρωτική σήμερα. Η στρατηγική για την κρίση δημιουργεί συγκεντροποίηση της πολιτικής. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Τι λέτε εσείς. Και πρόταση στην εισηγήτρια. Όταν μιλάτε για το εθνικό και περιφερειακό επίπεδο χρειάζεται να προσθέσετε και το τοπικό. Γιατί κάπου στην έκθεση μιλάτε για τοπικές επενδύσεις. Τοπικό δεν σημαίνει μικρός δήμος, Μπορεί να αναφέρεται και στο Παρίσι, το Λονδίνο, την Νάπολη κλπ. Γι' αυτό το τοπικό επίπεδο εν προκειμένου πρέπει να συμπεριληφθεί γιατί είναι σημαντικό. Πείτε μας λοιπόν τη γνώμη σας για αυτό το θέμα, συγκεντροποίηση έναντι εξυγίανσης και πώς θα είναι η πολιτική συνοχή στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο Βλάντιμιρ Μάγκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αρχικά δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά άκουσα τους εμπειρογνώμονες και αποφάσισα να πω και εγώ τη γνώμη μου. Επιτρέψτε μου καταρχάς να πω το εξής. Όλοι Συμφωνούμε ότι η πολιτική συνοχή και τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν σημαντικό μέσο στη μάχη κατά της κρίσης. Και στη Σλοβακία μέχρι 70% των δημοσίων επενδύσεων λαμβάνουν χώρα μόνο χάρη στα διαρθρωτικά ταμεία και χάρη στην πολιτική συνοχή. Η χώρα μας σήμερα έχει οικονομική ανάπτυξη, μικρή μεν, αλλά έχει χάρη, το ξαναλέω, στην πολιτική συνοχή. Οι εμπειρογνώμονες είπαν πολλά ενδιαφέροντα. Ένα ενδιαφέρον ε, ήταν αυτό που είπαν για τις υποδομές. Οι υποδομές δεν είναι πια ε, μοχλός ανάπτυξης. Είμαι και πρόεδρος μιας περιφέρειας, περιφερειάρχης στην Σλοβακία και έχω εποπτεία του χώρου. Στον τομέα της ενέργειας διαπίστωσα ότι αν επενδύσω στη θερμότητα, τότε μέσα σε τρία χρόνια έχω απόδοση της επένδυσής μου. Δηλαδή την παίρνω πίσω. Είναι καλή επένδυση και τα χρήματα που θα πάρω πίσω θα τα επενδύσω πάλι στην ανάπτυξη. Ε, χρήματα στις βασικές υποδομές μπορούν να επενδυθούν αλλά πρέπει να ε, επενδυθούν προσεκτικά και το ίδιο ισχύει και ε, για τις επενδύσεις ε, στην οδοποιία. Στα παλιότερα κράτη-μέλη τίθεται μεταξύ το ερώτημα γιατί να επενδύσει κανείς σε βασικές υποδομές όταν μπορεί να επενδύσει σε καινοτομίες. Σωστό και αυτό. Αλλά όταν ε, δεν επενδύουμε σε αυτοκινητόδρομους, σε δρόμους, τότε δεν θα έρθουν επενδυτές και θα στομώσουν οι περαιτέρω επενδύσεις και η ανάπτυξη. Εγώ στην περιφέρειά μου έκανα επενδύσεις στην οδοπία και τα χρήματα, είδα ότι τα χρήματα που μου υποσχέθηκαν από τα ταμεία δεν ήρθαν έγκαιρα. Το είδα και αυτό. Και όταν δεν γίνονται οι πληρωμές στην ώρα τους, τότε καθυστερούν και οι επόμενες επενδύσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το... Μην το ξεχνάμε και κατά την επόμενη περίοδο, την επταετή για τις επενδύσεις. Τα υπεσχημένα θα πρέπει να τηρούνται και οι πληρωμές πρέπει να γίνονται. Επί 8 χρόνια ήμουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και ε, κάποια στιγμή είχε γίνει ακρόαση της Επιτροπής η οποία ήθελε το 10% των επενδύσεων ε, να το ε, απαλείψει από τα νέα κράτη-μέλη. Γιατί τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούσαν να ε, απορροφούν έγκαιρα τα χρήματα. Αλήθεια ήταν αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως έβλεπα και στο δικό μου, στη δικιά μου τη χώρα την τεράστια γραφειοκρατία που φρενάρε τις επενδύσεις. Στη χώρα μου συνέβαινε αυτό. Η Κομισιόν ε, έλυσε πολλά προβλήματα, δηλαδή κατήργησε μεγάλο κομμάτι της γραφειοκρατίας και ευχαριστώ γι' αυτό, ήταν πολύ καλό. Τώρα όμως πρέπει να σκεφτούμε ε, και κάτι ακόμα. Δηλαδή θα πρέπει να ρωτήσουμε τις ίδιες τις περιφέρειες ποια έργα θέλουν και ε, για ποια έργα μπορούν να βρουν συγχρηματοδότηση, επενδύσεις. Υπενθυμίζω την προηγούμενη θητεία ε, τότε ήμουν εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2010. Και τότε στο Ευρωκοινοβούλιο είχαμε εγκρίνει ε, ένα σχέδιο για οικονομική έκθεση δύο γενικών διευθύνσεων για την ασφάλεια και την Ρέτζιο. Ε, Μία γενική διεύθυνση είχε μειώσει πολύ τις διοικητικές δαπάνες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ήθελε να κάνει και παρόμοια οικονομική εξέταση έρευνα και για το ίδιο το Κοινοβούλιο. Η οικονομική αυτή όμως εξέταση για το Κοινοβούλιο δεν έγινε. Πάντως και εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο μπορούμε να ε, προβούμε σε πολλές εξοικονομήσεις και να κάνουμε επενδύσεις πιο δυναμικές. Κάτι άλλο σημαντικό. Σε πολλά κράτη-μέλη τώρα ε, θεσπίζεται νομοθεσία που σκοπό έχει να φρενάρει το χρέος. Και στη Σλοβακία έχουμε περάσει παρόμοια νομοθεσία που είναι σημαντική πολύ. Αλλά και εδώ πρέπει να μην παραγνωρίζουμε κάτι σημαντικό. Ότι δηλαδή ορισμένες επενδύσεις έχουν ε, μέσα σε λίγους μήνες απόδοση. Αυτές οι επενδύσεις ε, όμως μπορεί να περιοριστούν από τις πολιτικές μείωσης και ανάσχεσης του χρέους. Ε, και μπορεί με την πολιτική μείωση ή ανάσχεση του χρέους να περιοριστούν αυτές οι θετικές πολιτικές. Δεν μπορούμε επίσης, όπως είπαν και οι ε, ειδικοί, να αυξάνουμε τη φορολογία ε, αυθαίρετα στα κράτη-μέλη για να μειώνουμε τα ελλείμματα. Αλήθεια είναι αυτό. Μην ξεχνάμε όμως ότι πριν από λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πέρασε νομοθεσία κατά των φορολογικών οάσεων. Υπάρχουν χώρες με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, χαμηλούς, άλλοι είναι παράδεισοι οάσεις που συγκεντρώνουν πολλά χρήματα. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ούτω ώστε να υπάρξει ένας αναπροσανατολισμός αυτών των φορολογικών οάσεων. Να μην έχουν χαμηλότερους ε, φορολογικούς συντελεστές αυτές οι οάσεις, αλλά να έχουν πιο φυσιολογικούς ή σε φορολογικούς συντελεστές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ε, αυτή είναι μια έκθεση την οποία θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε μέσα στα πλαίσια της αναζήτησης μιας ε, ευελιξίας στα πλαίσια της μακροαιρεσιμότητας και της ευελιξίας μεταξύ του μακροοικονομικού πλαισίου, στα πλαίσια του μακροοικονομικού πλαισίου. Θα ήθελα λοιπόν να ε, ρωτήσω, να ζητήσω από την εισηγήτρια να χρησιμοποιηθούν όλα τα πλαίσια ευελιξίας στα πλαίσια του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας έτσι ώστε στα πλαίσια των ε, μέσων που διαθέτουμε να δούμε πώς μπορεί να ενταχθεί η ευελιξία και πώς μπορούν να γίνουν αυτές οι, οι, οι, οι καταμετρήσεις για τις χώρες. Είμαι σχετικά ικανοποιημένος με τα νέα μέσα που δημιούργησε η ΕΤΕ. διότι οι δημόσιες αρχές δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα και γι' αυτό οι τράπεζες πρέπει να ε, συμμετάσχουν και να συμμετέχουν γενικότερα ε, ενεργά πώς οι εμπειρογνώμονες βλέπουν αυτά τα μέσα που έχει δημιουργήσει η ΕΤΕ έτσι ώστε να υπάρχουν εγγυήσεις και από την ΕΤΕ και ε, στα πλαίσια των δικών μας ταμείων, έτσι ώστε να έχουμε συνεχείς ε, ροές στην ε, χρηματοπιστωτική αγορά. Γιατί να μην μπορούμε να ε, γιατί να μπορούμε να προσμετρήσουμε και αυτές τις επενδύσεις, διότι αυτές είναι βιώσιμες, αυτές ελέγχει η και ούτω καθεξής. Αυτά είναι παραδείγματα. Γιατί ακριβώς μιλάμε όταν μιλάμε για ευελιξία. Θα ήθελα να το ψηφίσουμε αυτό και να το θέσουμε στην Ολομέλεια. Θα πρέπει στο δεύτερο ε, εξάμεινο του έτους να ε, ορίσουμε επακριβώς και τους ε, δικούς μας ε, κανονισμούς στα πλαίσια μιας δημόσιας συζήτησης και βεβαίως είμαστε και υπόλογοι ενώπιον των εκλογέων μας του χρόνου. Ευχαριστώ Λαμπέρ Φραντσέσκο Ντε Ευχαριστώ Πρόεδρε κατανοώ απόλυτα τη θέση της εισηγήτριας και συμμερίζομαι τα ε, σχόλιά της σε σχέση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του ε, Ιουλίου του 12 και των αρχών του 13 σε σχέση με τα δημοσιονομικά. Πρόκειται για ένα δυσμενές έτος διότι οι περιφερειακές ανισότητες αυξάνονται ανά την Ευρώπη παρά την πολιτική συνοχής που προϋπάρχει. Εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη την περίοδο 2014-2020, στα πλαίσια των δυσχεριών και της ε, κρίσης, αυτά είναι και τα μοναδικά μας μέσα για να προωθήσουμε την ε, ανάπτυξη στα πλαίσια της δυνατότητας χρηματοδότησης ε, νέων προγραμμάτων για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και γενικότερα την εργασία. Σε μια στιγμή μεγάλων ε, δυσχεριών και στα πλαίσια της πολιτικής λιτότητας. Σημερίζομαι τους στόχους της στρατηγικής 2020 στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης που μπορούν να συμμεριστούν και οι τοπικές αρχές, τη διαφάνεια στη δημοσιονομική διαδικασία και τον, την αναγνώριση των μέσων χρηματοδότησης. Επίσης θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε αυτές τις πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις πολιτικές χρηματοδότησης, γιατί δεν μπορούν να οριστούν παρά στα πλαίσια μίας συμμετοχής των τοπικών αρχών. Μιλάμε για την πρόθεση της ανάπτυξης. Ποιοι θα είναι οι, οι πόροι μας όμως, ποια θα είναι τα μέσα μας. Είμαστε πεπισμένοι για αυτή την ανάπτυξη, αλλά όχι για τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους και τα μέσα. Και να δούμε πώς θα ορίσουμε τις εθνικές επενδύσεις. Να μας απασχολήσει και η συγχρηματοδότηση, διότι πολλές φορές δεν υπάρχει ευελιξία στα πλαίσια της χρήσης του Συμφώνου Σταθερότητας. Πώς μπορεί να οριστεί επακριβώς η συγχρηματοδότηση που πολλές φορές ε, μπλοκάρει την εισρωή πόρων, ιδιαίτερα στις μειονεκτούσες περιοχές. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε και ένα άλλο θέμα που αφορά την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Διότι συζητήσαμε αυτό το ζήτημα, όλες οι ομάδες έχουν εκφράσει, έχουν εκφραστεί ως προς το γεγονός των δημόσιων, ως προς τα δαπάνες αυτό το είδαμε και στη Ρέτζη μέσω τριμερών διαλόγων. Όμως οι διαθεσμικές διαπραγματεύσεις επιβεβαιώνουν την αιρεσιμότητα και γι' αυτό θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το σημείο. Πώς δηλαδή οι συζητήσεις μας και η έγκριση αυτού του πλαισίου θα οδηγήσει σε επιτυχία των τριμερών διαλόγων ως προς τον μελλοντικό προγραμματισμό της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Να προσθέσω μία παρατήρηση γιατί πολλές φορές ξεχνούμε από πού παίρνουν τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανεπτύξεως επενδύσεων, συγγνώμη. Παίρνει τα χρήματα από εκεί που παίρνουν και άλλε τράπεζε. Και οπότε γι' αυτό το λόγο και πολλέ φορέ κοντράρονται μεταξύ του. Ε, οπότε <laughs> ακριβώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό είναι το, το, το πρότυπο. Δεν έχουν κάποια άλλη συνταγή. Τώρα παρακαλώ οι καθηγητέ, αν θέλουν, μπορούν να, να δευτερολογήσουν. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, ε, ό,τι θέλετε. Και μετά στη συνέχεια η κυρία Ματσόνη μπορεί επίση να κλείσει τη συζήτηση. Αλλά πρώτα-πρώτα η προσκεκλημένη μα υπάρχουν πολλές, πολλές παρατηρήσεις, να είμαι σύντομος, διότι δεν θέλω να σας μιλήσω για την ε, ε γραφειοκρατία μόνο, αλλά τι να σας πω, πάτε στο Στασβούργο και πηγαίνω έρχεστε εκεί πέρα. Έτσι αυτό το λέω για κάποιο τρόπο έτσι περιπεκτικά προς εσάς, αλλά τι θα γίνει με αυτή τη συνδιαχείριση. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, πολλά χρόνια δούλεψα για τέτοιες υποθέσεις σαν σύμβουλος, σαν πανεπιστημιακός, από όλε τι επόμενε οπτικές γωνίες έχω αντιμετωπίσει το θέμα. Μπορώ να σας πω, σε σχέση με τη διαμόρφωση των στρατηγικών που έχω τόσο πολύ ζήσει, ότι είναι ότι έχουμε προγράμματα τα οποία έχουν χαραχθεί, ε, η διαχείριση τους γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Έτσι σχεδιάστηκαν όμως. Θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα καλά. Και αυτό είναι και το θέμα. Γιατί έχω δει πάρα πολύ κακό προγραμματισμό αλλού, αλλού πάρα πολύ καλό. Ε, με αυτό ακριβώς είναι και το θέμα. Και βέβαια, όποιος ε, βλέπει, άλλος βλέπει μισογεμάτο ποτήρι, άλλος μισοάδιο, αλλά τέλος πάντων όταν εγώ ξεκίνησα τη διαδρομή μου για τα θέματα τα δημοσιονομικά, τότε το, το, το, ήταν τα ερωτήματα απλά. Έχουμε 50% ή 30% συγχρηματοδότηση, θα πληρώσουμε ή θα πληρώσουμε για τις αγελάδες. Τώρα όμως ε, φτάσαμε να μιλούμε για χρηματιστηριακά προϊόντα, για εγγυήσεις, για θέματα που πριν από 15 χρόνια κανένας κανένας δεν είχε κάτι να πει. Οπότε φτάνουμε τώρα σε αυτή την ε, ε, τεχνική αρρωγή. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τη διοίκηση. Αφορά και τις τράπεζες. Γιατί η ΕΤΕ μέσω των τραπεζών ρίχνει πολλά χρήματα στο σύστημα. Οπότε βλέπετε ότι καμιά φορά δεν μπορεί ο τραπεζικός τομέας να κρατήσει τον ρυθμό. Η EBRD, η Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τι κάνει. Εκπαιδεύει ούτως πίν. έχει πολύ στενή επαφή με αυτές τις τραπεζικές κινήσεις που σας ανέφερα. Και πολλές φορές όμως οι τράπεζες δεν είναι προετοιμασμένες. Δεν έχουν την ούτως πίν τεχνογνωσία, την εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζεται. Άρα θα πρέπει να προβληματιστούμε πώς θα βοηθήσουμε, πώς θα παρακολουθήσουμε την επιλογή των προγραμμάτων, να δούμε τι γίνεται στο τοπικό επίπεδο. Δεν μιλώ για παρέμβαση, μιλώ για βοήθεια, μιλώ για παρακολούθηση. Ε, δεν μπορεί κανείς να μην βοηθάει τις χώρες και μετά να τις επικρίνει γιατί δεν τα κατάφεραν καλά. Επομένως, θα πρέπει κανείς να προβληματιστεί γιατί θα πρέπει να δούμε αν για την επόμενη περίοδο και τον προγραμματισμό τη, αν θα έχουμε στρατηγική ικανότητα στο τοπικό επίπεδο. Κάτι το οποίο δεν απέδωσε στο παρελθόν για τα απλά προγράμματα. Ε, άρα τώρα κατά μείζον λόγο για τα πιο περίπλοκα θα πρέπει να σκεφτούμε, να προγραμματιστούμε περισσότερο. Επίση, για την προσθετικότητα και την απορροφητικότητα. Αυτό που έχει σημασία βέβαια είναι η των στόχων. δεν διαπίστωσα να υπάρχει μετά από 7 χρόνια εάν για κάποιο πρόγραμμα εάν κανείς ασχολήθηκε με το αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Όλοι ασχολούνται με την απορροφητικότητα. Εάν κανείς δεν ασχολείται με αυτό, πώς να πετύχει τους στόχους. Άρα τόσο θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποιους ξεκάθαρους δείκτες, κριτήρια, πώς θα υπάρχει η παρακολούθηση. Γι' αυτό και σας μιλώ για βοήθεια και για παρεμβατική τακτική. Δηλαδή κανείς να είναι παρόν και να ακολουθεί τους δείκτες τα κριτήρια. Λίγα είναι αυτά τα κριτήρια και ξεκάθαρα. Για την προσθετικότητα τώρα υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Το καταλάβαινα στο παρελθόν, γιατί όλοι ήταν πλούσιοι. Παντού υπήρχε ανάπτυξη και προσθετικότητα σήμαινε ότι κανείς θα προσθέσει, θα, θα, θα ξοδέψει το, ίδιο ποσό και κατόπιν θα τα πάρει πίσω. Και δεν υπήρχε καν πραγματικός έλεγχος εάν τα χρήματα πήγαιναν τυχόν κάπου άλλο, αλλού. Θα πρέπει τώρα στην κρίση να πούμε σε κάθε χώρα ότι θα πρέπει να κόψει κατά πολύ τις δημόσιες δαπάνες και μετά όμως λέμε στις χώρες δεν θα πάρετε το κοινοτικό χρήμα, την κοινωνική ενίσχυση, εάν δεν υπάρχει η προσθετικότητα. Αυτό άρα σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα λογικής αντίφασης εδώ. Χρειάζεται η υποδομή, χρειάζεται για την ανάπτυξη, όμως δεν είναι η μόνη προϋπόθεση για να φτάσουμε την ανάπτυξη. Η Σλοβακία καλά τα πάει με την υποδομή, αλλά άλλοι όχι τόσο καλά. Και πολύ σημαντικό βέβαια είναι ο προγραμματισμό για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το καλό είναι ότι η ΕΤΕ έχει μια κατάταξη βαθμολόγηση. Επομένως είναι πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά την ποιότητα των προγραμμάτων. Το κακό ποιο είναι τώρα. Υπάρχει πρόβλημα εδώ με το ρίσκο. Εκεί που υπάρχει ρίσκο δεν τολμούν να ασχοληθούν. Για την Ελλάδα, ξέρω εγώ, για να τη βοηθήσουν να βγει από το αδιέξοδο. Ε, φοβούνται, φοβούνται εκεί πέρα να ασχοληθούν. Για τη γενοτομία, ας πούμε. Με εξέπληξε ότι μετά από τόσα χρόνια δεν υπήρξε κανένα πρόγραμμα το οποίο να κατέρευσε. Άρα, να έχουμε κίνδυνο 20% να, από, καταρρεύσουν τα προγράμματα, ε, να μην έχει καταρρεύσει κανένα. Άρα τότε γιατί κανείς να φοβάται να ρισκάρει, αφού μια χαρά πήγαν τα προγράμματα. Αυτά και τώρα δίνω στο κοιτάλι στον παρακαθήμενο. Ευχαριστώ και πολλά και εύστοχα σχόλια ετέθησαν. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα μέσα που έχουμε για την πολιτική συνοχή ε, πληρούν το χάσμα ε, σε σχέση με μειονεκτούσες και αναπτυγμένες περιοχές, δηλαδή κατά πόσο είναι θέμα λιγότερων ε, ή περισσότερων πόρων ή θέμα απορροφητικότητας. Ε, το δεύτερο ερώτημα που έθεσε η κυρία Ματσόνη είναι ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για μία εξαίρεση ως προς το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι επιπτώσεις είναι ουσιαστικές ή όχι. Θα πρέπει να γίνει μία πιλωτική έρευνα για να δούμε κατά πόσο η συλλογιστική αυτή της ε, δημοσιονομικής λιτότητας είναι αποδοτική. Ε, δεν συμφωνώ με τον κύριο Όλμπραϊτ. Χρειάζονται χρειάζεται να ξεπεράσουμε αυτό τον δημοσιονομικό γόρδιο δεσμό για να επιτύχουν οι πολιτικές μας, αλλά υπάρχει και χρηστή διαχείριση. Θα ήθελα να μπορώ να συμμεριστώ τις απόψεις του συναδέλφου μου όταν μιλάμε για τις τοπικές αρχές και την αυτόνομη δράση τους. Όταν μιλάμε για εθνικές στοχοθετήσεις θα πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο μπορούμε να άρουμε αυτό το, τον ε, δημοσιονομικό βρόχο και παράλληλα να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να εξηγιανθεί η δημοσιονομική κατάσταση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Βεβαίως, τίθεται και θέμα διαχείρισης μέσα στα πλαίσια μιας εθνικής στρατηγικής. Συμφωνούμε με αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει χρηστότερη διαχείριση. Διαφορετικά θα ήταν άκρος απογοητευτικό το όλο εγχείρημα. Υπ' αυτή την έννοια δεν έχει νόημα να προβλέπουμε μόνο κυρωτικούς μηχανισμούς θα πρέπει να αναπτύξουμε προγράμματα, όχι να θέτουμε, ε, να επιβάλλουμε κυρώσεις σε προγράμματα τα οποία δεν αποδίδουν. για να ενδυναμώσουμε την ευελιξία, για να ενισχύσουμε την ευελιξία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλαπλούς παράγοντες εγώ κινούμαι στην Ευρώπη εδώ και μακρύ χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θέτουμε τη συγχρηματοδότηση εκτός συμφώνου σταθερότητας ή όχι. Γιατί ορισμένες ε, συμφωνίες έχουν ήδη ληφθεί ενδοκινοτικά. Εάν όμως γίνουν δαπάνες όπου εμπεριέχονται οι φόροι που επανέρχονται στο κράτος, γιατί, γιατί να μην ε, εμπεριέχονται στην εθνική ε, λογιστική, στο εθνικό λογιστικό σύστημα δηλαδή σε ένα 40 επί με ενδιαφέρει κατά πόσο εμπεριέχεται ο ΦΠΑ, ο οποίος είναι της τάξης του 8 ή 9% και κατά πόσο εντάσσεται στην εθνική, στα εθνικά λογιστικά βιβλία. Θα πρέπει να είμαστε πιο συνεκτικοί, λοιπόν. Γιατί δεν μπορούν αυτά να ενταχθούν στην πολιτική συνοχής. Γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε όμως τους φόρους από τις εθνικές ή τις δημόσιες αυτές δαπάνες. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, και την φορολόγηση μέσα στα πλαίσια της ε, ε, λογικής, της παραγωγικής αυτής λογικής ερμήνεια. Θα είμαι πολύ σύντομη Οπωσδήποτε θα λάβω υπόψη τις συνεισφορές όλων. Ε, εφήγησαν πολλά και σημαντικά ζητήματα. Λαμβάνω υπόψη και τις αντιρρήσεις που προέβαλαν μερικοί. Οι δύο μας, οι εμπειρογνώμονες απάντησαν επαρκώς και δεν χρειάζεται να προβάλλουμε και άλλα στοιχεία. Εδώ ε, αναφέρομαι στα, όσα προανέφερε και ο συνάδελφος Γκοντμάνης, ο οποίος με πάθος επέκρινε την βασική συλλογιστική της έκθεσης και έθεσε μια σειρά ερωτημάτων σε σχέση με το θέμα της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Μας ενδιαφέρει η απόδοση, η αποδοτικότητα της επενδυτικής μας πολιτικής και νομίζω ότι και ο ε, καθηγητής ε, Μουστήλη απάντησε και ο καθηγητής Φερέρ μας ε, προέβαλε μία επιχειρηματολογία μιλώντας για την αποδοτικότητα ή μη του συστήματος. Βεβαίως, εμείς δεν παράγουμε και γι' αυτό δεν είναι και λειτουργικό το σύστημα. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να εξεύρουμε και διαφορετικές λύσεις από αυτές που προτείνω εγώ. Θα πρέπει όμως να προταθούν. Ως προς το ερώτημα του κυρίου Όλμπριχτ, νομίζω ότι εδώ ε, δόθη απάντηση από τους δύο καθηγητές Μας ενδιαφέρει να δούμε και το θέμα αυτού του συγκεντρωτισμού των πολιτικών μας και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει ο τοπικός παράγων να ε, δράσει άμεσα. Μέσα στα πλαίσια της νέας μας ατζέντας προτεραιοτήτων για να δούμε πώς ε, μπορούμε να έχουμε αθρώα τοπική συμμετοχή. Συμμετοχή από τις τοπικές αρχές δηλαδή για την ε, υλοποίηση της ε, πολιτικής συνοχής. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να εντάξουμε σε μία συλλογιστική εθνικής στρατηγικής διότι πρέπει να δράσουμε μέσα στα πλαίσια μιας αναπτυξιακής πολιτικής που να ενταχθεί και να συνδέεται με τα μέσα συνοχής που διαθέτουμε προσπαθώντας να άρουμε τα προσκόμματα που προϋπάρχουν. Ως προς το ερώτημα του κυρίου Βανίστελ Ρόι, για το σημείο 13, νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα μέσα και δυνατότητες ευελιξίας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μας δώσει απαντήσεις. Μιλήσαμε για, τον, ε, για τη φορολόγηση και τον υπολογισμό των φόρων, όπως μας ε, είπε ο καθηγητής μου Στήλη. Αυτά είναι ένα από τα μέσα, μία από τις υποθέσεις εργασίας για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις ε, δημοσιονομικές προσταγές και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας επενδύσεων. Ως προς την παρέμβαση De Angelis, όπως είπα, ε, ως προς την μακροαιρεσιμότητα έχουν ε, υποθεί πολλά. Και πιστεύω ότι όλες οι υποδείξεις είναι χρήσιμες και θα τις λάβω πολύ σοβαρά υπόψη. Μπορούμε να εμπλουτίσουμε το έγγραφο και με τροπολογίες. Θα ήθελα να ρωτήσω την Προεδρία ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα γιατί δεν το γνωρίζω. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες στην Κομισιόν, τους συνάδελφους που πήραν το λόγο σε αυτή την τόσο χρήσιμη συζήτηση. Ευχαριστώ και την κυρία Ματσόνη που μας έδωσε την ευκαιρία για τη συζήτηση αυτή. Η μόνη απόφαση είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών μέχρι 4 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Ελπίζω ότι θα ψηφιστεί τον Ιούλιο. Αν λόγω των ψηφοφοριών του Ιουλίου δεν προλάβουμε, θα πάει Σεπτέμβρη. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα τα καταφέρουμε όλα αυτά. Κατά βάση μπορεί να γίνει τον Ιούλιο. Θα εμείς θα προσπαθήσουμε να περάσει τον Ιούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τώρα τη συζήτηση. Τώρα έχουμε από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο συναδέλφους εδώ, την κυρία Γκάφη. Θα μιλήσουμε για την ε, έκθεση στρατηγικής και την εφαρμογή στην ε, τωρινή περίοδο, προγραμματική περίοδο των προγραμμάτων. Βερόνικα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέω να, κάνουμε, να κάνω μια παρουσίαση και μετά να ακολουθήσει η συζήτηση. Μέχρι τώρα που ετοιμάζεται η οθόνη θέλω να σας πω ότι θα παρουσιάσω τη δεύτερη έκθεση στρατηγικής 2017-2013. Ε, την πρώτη την παρουσιάσαμε το 2010 μαζί με τον Τζον Walsh Ελπίζω να καταφέρομαι να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας και με ενδιαφέρον θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις σας στην έκθεση. Η έκθεση 2013 στηρίζεται σε 27 εθνικές στρατηγικές εκθέσεις σε 2.000 σελίδες ανάλυση του τι πέτυχε μέχρι τώρα η πολιτική συνοχή στην τωρινή προγραμματική περίοδο και ποια είναι τα κέρια μηνύματα της έκθεσης. Η πολιτική συνοχή συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και στις θέσεις εργασίας και τους στόχους που έχουν τεθεί. Αναφέρομαι σε αυτό το προηγούμενο που ελέγχθη ότι κανείς δεν κοιτάει αν επιτυγχάνονται οι στόχοι. Εμείς τα κοιτάμε αυτά και ελπίζουμε να εντείνουμε την εστίαση αυτή στην επίτευξη των στόχων. Η υλοποίηση αυξήθηκε, έχουμε σημαντικά αποτελέσματα σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Η Κομισιόν ε, δείξε ότι έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε αλλαγέ ε, αναγκών. Τώρα περιμένουμε πολλά αποτελέσματα και στην τωρινή σημαντικά στην ε, προγραμματική περίοδο πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες και να δούμε αυξημένους κινδύνους που υπάρχουν σε κάποιους τομείς και κράτη-μέλη. Για να δούμε λοιπόν τώρα ε, ποια είναι ποιος είναι ο αντίκτυπος της ε, κρίσης. το σοκ διαφέρει ως προς την σοβαρότητά του. Μια, στρατηγική, μια έκθεση στρατηγικής έδειξε ότι αναδείχθηκαν προτέρες αδυναμίες ε, είδαμε λοιπόν ποια, ποιον αντίκτυπο είχε η κρίση στις διάφορες χώρες. Υπάρχουν διαφορές σχετικά με την εκτίμηση της πολιτικής συνοχής. Στα βόρεια κράτη-μέλη ε, έχουμε θέμα Ε, ε, εκεί η στρατηγική συνοχή είναι στρατηγική πλατφόρμα σημαντική και η στρατηγική που αναπτύχθηκε στην αρχή της περίοδου ε, εξακολουθεί να είναι σημαντική. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 12 βλέπουμε διαφορετικά να έχει αντίκτυπο η κρίση αλλά το βασικό είναι ότι θα πρέπει να δούμε τα το μέγεθος των προγραμμάτων που έχει διαφοροποιηθεί. Για τα νότια κράτη-μέλη βλέπουμε ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες κυριαρχούν και η πολιτική συνοχή θεωρείται σημαντική υποστήριξη των επενδύσεων. Υπάρχουν ε, δείγματα αυξανόμενων περιφερειακών ανισορροπιών με την κρίση όμως. Ποια ήταν η απάντηση. Καταρχήν βλέπουμε ότι υπάρχει μειωμένη ζήτηση και στήριξη της Ένωσης σε πολλούς τομείς ε, καινοτομίες ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε μακρότερες περιόδους παράδοσης, επιβράδυνση ε, της ε, ε, ε ικανοτήτων ε, προβλήματα στην πρόσβαση, στην χρηματοδότηση, υποδομές, ε, έρευνας, ανάπτυξης, τεχνολογίας. Βλέπουμε σημαντικό στρες στην ικανότητα ε, της διοίκησης να ανταποκριθεί στα παραδοτέα. αυτό είναι μια πρόκληση σε ορισμένες ε, περιπτώσεις. Και υπάρχουν αβεβαιότητες και προβλήματα σε σχέση με τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις και τα, τα προγράμματα λιτότητας. Για να δούμε την απάντηση λοιπόν. Υπάρχουν μέτρα κατά της κρίσης, τα οποία έλαβε η Κομισιόν, ε, προκαταβολές, ε, επιτάχυνση μεγάλων προγραμμάτων, απλοποίηση και κάναμε αναπρογραμματισμό της συγχρηματοδότησης. Αν δούμε τώρα τον αναπρογραμματισμό της θεματολογίας, 35,7 ε, δις ευρώ είχαν δοθεί ε, μεταξύ 86 θεμάτων ή κατηγοριών επενδύσεων που είναι 10,3% όλων των ε, κονδυλίων. 86% αυτών έγιναν το 2011-12. Από τότε που ολοκληρώσαμε την ανάλυση στην έκθεση στρατηγικής, ε, ο αναπρογραμματισμός θεματικών έφτασε στο 39,2 δις μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Οι περισσότερες αναδιανομές έγιναν από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ 30,2 δις και το κοινωνικό 5,5 δις. Ε, αυτός ο αναπρογραμματισμός είναι μεταφορές μέσα σε μεγάλα θεματικά, θεματικές ενότητες και μεταξύ θεματικών ενότητων. Αλλά αυτό διαφέρει, υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ κρατών μελών. Εδώ έχουμε μία σύνοψη όλων των ποσών αυτό που βλέπουμε είναι ότι η πολιτική έχει την ικανότητα να είναι αρκετά ευέλικτη για να προσαρμόζεται σε κρίσεις. Έγινε αναπρογραμματισμός της συγχρηματοδότησης με μείωση της εθνικής συμμετοχής. Το σημείο εκκινήσεως όταν άρχισαν τα προγράμματα ήταν 347 δις ε, κοινοτικής χρηματοδότησης και 133 εθνική χρηματοδότηση. Η εθνική χρηματοδότηση έπεσε στα 126 δις στο τέλος του 2012, μειώθηκε κατά 15 δις και επικεντρώνεται σε κάποια συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι θα γίνονται κάποιες επενδύσεις, σημαντικές επενδύσεις να γίνονται. Αναγνωρίζουμε όμως ότι μειώνουμε τη συνολική προσπάθεια και αυτό έχει επιπτώσεις σε σχέση με την προσθετικότητα. Όμως η γνώμη της Κομισιόν ήταν ότι χρειαζόταν ανάληψη κάποιας δράσης λόγω της πρωτόγνωρης κρίσης. Για να δούμε τώρα το ημείωση των συντελεστών της εθνικής χρηματοδότησης, συγχρηματοδότησης που επικεντρώνεται. Επικεντρώνεται στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λατωνία, Λιθουανία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Όλα τα προγράμματα, δηλαδή ε, χωρών που επλήγησαν πολύ από την κρίση συμβολή στο Ευρώπη 2020. Στις εκθέσεις τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν τη σημασία της πολιτικής συνοχής που στηρίζει ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλους τους τομείς. Τώρα το εγχείρημα της Λισαβόνας για τη δέσμευση χρημάτων του 2007 εξακολουθεί να ισχύει με τους πυλώνες, ε, τους ε, έξυπνους και τους ε, χωρίς αποκλεισμούς. Τώρα για το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη, πολλές εκθέσεις αναφέρθηκαν στο Σύμφωνο και τη σημασία της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες όπου η πολιτική συνοχής και οι επενδύσεις μέσα από εκεί είναι η μόνη επένδυση που λαμβάνει η χώρα στις χώρες αυτές. Αλλά πρέπει να δούμε τις 27 ε, εκθέσεις στρατηγικής για να πάρουν πιο πολλές πληροφορίες εδώ. Εδώ είναι τα καινούργια κομμάτια όπου μπορούμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τις αποδείξεις αποτελεσματικότητας και επιδόσεων. Το βασικό μήνυμα είναι ότι βλέπουμε σημαντικές αυξήσεις ε, στην, ε, στα αποτελέσματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια μεγάλη συμμετοχή στην εκπαίδευση και ανακατάρτιση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ενδιάμεσες πληρωμές που δηλώθηκαν είναι 42% των πιστώσεων που ήταν διαθέσιμες τέλος Ιανουαρίου. Τώρα έχουμε πάει στο 45%. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα έχουμε πολλή υλοποίηση να κάνουμε τώρα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Η επιλογή των έργων ε, είναι σημαντική στα πλαίσια των επιδόσεων γιατί πρέπει να δούμε τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες που ε, διοχέτευσαν τα χρήματα, ποια έργα επέλεξαν. Στο τέλος του 2011 είμαστε στο 71% των διαθέσιμων πόρων και υπολογίζουμε 88% στο τέλος του 2012. Λοιπόν, εδώ τώρα μιλάμε περισσότερο για την ανάγκη να πάμε πέρα από την απορροφητικότητα και να δούμε τι έχει επιτευχθεί μετά την δαπάνη των χρημάτων αυτών. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στις εκθέσεις στρατηγικής, στην έκθεση στρατηγική στη δικιά μας είναι ότι ε, έχουμε ε, ε, φύλλα παρακολούθησης δικτών, βλέπουμε τι έγινε, βασικούς δείκτες και συγκρίνουμε με την επιλογή των έργων και την απορρόφηση των κονδυλίων και αναλύουμε τα αποτελέσματα. Το βασικό, ε, αυτά, αυτοί είναι οι βασικοί δείκτες. Αυτά μπορούμε να τα παρουσιάσουμε συγκεντρωτικά σε ενωσιακό επίπεδο. Ε, όλα αυτά που γίνονται ε, δεν είναι, περιλαμβάνονται βέβαια, είναι πολλά τα δεδομένα που βλέπετε και οι λεπτομέρειες στις εκθέσεις στρατηγικής, στις εθνικές. Ε, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό είναι κάτι που διαπραγματευτήκαμε και συμφωνήσαμε με τα κράτη-μέλη, αλλά δεν προβλέπεται από τον κανονισμό για την τρέχουσα περίοδο. Η χρήση κοινών δικτών για την επόμενη προγραμματική περίοδο όμω θα καταστεί υποχρεωτική. Αυτό που κάνουμε λοιπόν στην τωρινή προγραμματική περίοδο είναι σε εταιρική σχέση, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, να πτήσουμε την ικανότητα να παρακολουθούμε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ε, για να μπορούμε να ε, έχουμε καλά στοιχεία όχι μόνο για την απορροφητικότητα και την καλή ε, χρήση των πόρων αλλά και τα αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν σημαντική επιτάχυνση της προόδου σε σχέση με τους βασικούς δείκτες το 2011. Συνεχίζεται η καλή πορεία και το 2012. Ε, θέσεις εργασίας, 400.000 θέσεις εργασίας ε, δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2011. 15.000 είναι έρευνα ανάπτυξη και τεχνολογία και πολλές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, βλέπουμε ε, νεοσύστατες επιχειρήσεις να ε, στηρίζονται τα ευρυζωνικά μέσα πρόσβαση στα στα πόσιμο είδωρ, καλύτερη αποχέτευση, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Για να δούμε τώρα το στοιχείο για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν ε, είναι ε, τέλεια όλα. Αυτά τα ε, εξελίσσουμε και τα τελειοποιούμε μαζί με τα κράτη-μέλη και αναλύουμε τα δεδομένα, τα συζητούμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τις διαφορές στις αναφορές και εκθέσεις που παίρνουμε. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Γι' αυτό τα κάνουμε αυτά στις συζητήσεις μας για τις επιδόσεις των πολιτικών. Αν δούμε εδώ το πίνακα για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκε βλέπουμε κάποια παράδοξα που πρέπει να τα συζητήσουμε περισσότερο με τα κράτη-μέλη για να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει. Ε, η Δανία, για παράδειγμα, δεν αναφέρει δημιουργία θέσεων εργασίας. Γιατί? Διότι το 2007 στη Δανία η δημιουργία θέσεων εργασίας δεν φαινόταν να είναι νομίζων στόχος για τα διαρθρωτικά ταμεία. Ενδιαφέρονταν περισσότερο για την παραγωγικότητα, οπότε δεν το επέλεξαν αυτό ως δείκτη. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα που αφορούν ορισμούς, δεδομένα ε, κωδικοποιημένα, αλλά θα τα βελτιώσουμε αυτά ε, ε, στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περίοδος, περίοδου για να έχουμε καλύτερους δείκτες στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Τώρα, για τα έργα αυτά που δίνουμε σε σχέση με τις πληρωμές. 71% είναι ο μέσος όρος, μερικά είναι 100% αλλά είναι κάτω από 60% στα κρατη 42% του προϋπολογισμού ε, παρουσιάστηκε ως ενδιάμεση πληρωμή. Υπάρχει μεγάλη διακείμενση στις δαπάνες στα κράτη-μέλη και αν ε, μεταφράσουμε τα επιλεγμένα προγράμματα ε, σε δαπάνες και αυτό έχει διαφορές. Οπότε 32 ε, μήνες μένουν μέχρι το τέλος του 2015, 30 μήνες. Υπάρχουν αυξανόμενοι κίνδυνοι σε κάποια ότι οι δαπάνες δεν θα λάβουν χώρα και δεν θα ε, υπάρξουν ωφέλη. Για να δούμε εδώ ε, στην έκθεση στρατηγικής από τα κράτη-μέλη βλέπουμε την κατανομή των, των πόρων μέχρι το 2011 με μπλε το κόκκινο είναι οι πληρωμές που παρουσιάστηκαν, δηλώθηκαν στην Κομισιόν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Και βλέπουμε υψηλή απορρόφηση σε κάποια κράτη-μέλη, Αυστρία, Βελγίο, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σουηδία, αλλά έχουμε προβλήματα σε κάποια άλλα κράτη-μέλη. Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβακία και ιδιαίτερα νομίζω ε, στη Ρουμανία υπάρχουν προβλήματα. Οπότε εδώ βλέπετε το εύρος της πρόκλησης και τη διακύμανση στα κράτη-μέλη. Όμως, αν δούμε τις θεματικές τάσεις, γιατί αυτή είναι η συνολική εικόνα, τα δεδομένα από το τέλος του 2011 ε, ε, ε, είναι ηλικίες 17 μηνών. Δηλαδή περνάει χρόνος ε, μέχρι να φτάσουν σε εμάς τα στοιχεία. Ε, τέλος Ιουνίου του 2013 θα πάρουμε κι άλλα στοιχεία. Τέλος του επόμενου μήνα δηλαδή, οπότε θα πιάσουμε μέχρι το τέλος του 2012. Βλέπουμε όμως συνεχείς διαρθρωτικές καθυστερήσεις σε κάποια κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα μας απασχολεί το θέμα της ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές, ευρυζωνικά, δημιουργία ικανοτήτων ε, σιδηρόδρομοι βλέπουμε εδώ ε, υπό και υπερπρογραμματισμός που δεν φαίνεται πολύ μέχρι τώρα. Μπορεί να χρειαστεί αναπρογραμματισμός. Αυτό θα γίνει αργότερα στα πλαίσια της προγραμματικής περίοδου. Βλέπουμε εδώ την επιλογή των έργων για τις βασικές θεματικές ενότητες. Βλέπετε ότι η κόκκινη γραμμή είναι ο μέσος όρος και βλέπετε κάποιους τομείς που υπολείπονται, έρευνα, ανάπτυξη, IT, ε, ενέργεια, σιδηρόδρομοι, δημιουργία ικανοτήτων. Αν πάρω ένα θέμα, πάρουμε, πάρουμε τους σιδηροδρόμους. Ε, βλέπετε εδώ το, την, το, ταχύτητα επιλογής 60% που είναι κάτω από το μέσον όρο που είναι 70% για όλες τις θεματικές ενότητες και βλέπουμε ιδιαίτερα προβλήματα σε κάποια κρατημέλη, Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία, Λιθουανία, Σλοβενία. Εδώ αυτές διακρίνονται και δίνονται πολλά χρήματα σε κάποιες από αυτές, Πολωνία για παράδειγμα. Αυτή είναι η τομή όπου έχουμε πραγματικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Συμπεράσματα. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που πρέπει να βελτιωθούν ως προς την ταχύτητα επιλογής. Το 2012 και το 2013 το βλέπουμε αυτό. Και το βλέπουμε με βάση τα δεδομένα ε, που πήραμε και αυτά που θα πάρουμε Υπάρχουν κίνδυνοι σε ορισμένες θεματικές ενότητες και υπάρχει, χρειάζεται υψηλή εστίαση στην υλοποίηση των προγραμμάτων των τωρινών. Ε, πιέζουμε τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν τις προσπάθειες υλοποίησης των τωρινών προγραμμάτων και μην ξεχνάμε τα τωρινά προγράμματα και την προετοιμασία, μην ξεχνάμε τα τωρινά προετοιμάζοντας τα επόμενα. Ε, πολλά γίνανε, αλλά πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν. Τώρα, ε, τάσεις για το μέλλον, τελευταία μου διαφάνεια, για την τωρινή τρέχουσα περίοδο συμπεραίνουμε ότι υπάρχει δυναμική στην αναγνώριση της πολιτικής συνοχής και της σημασίας της, ιδιαίτερα στην κρίση, αυξάνει τη σημασία της, ε, αλλά πιο πολύ μεγάλη προσπάθεια υλοποίησης χρειάζεται και εξαίρενση μείωση της εθνικής συγχρηματοδότησης θα εξεταστεί όπου χρειάζεται, αλλά όταν στοχεύουμε υψηλής προτεραιότητας μίς και ε, όταν πραγματικά ε, στοχεύουμε στην ανάπτυξη. Για το μέλλον, κάποια κράτη-μέλη στις εκθέσεις στρατηγικής αντλούν διδάγματα για μελλοντικές προτεραιότητες και την ευελιξία στα πλαίσια της κρίσης. Εμείς ε, συμπεραίνουμε επίσης ότι υπάρχει ανάγκη αποφυγής καθυστερήσεων και ε, όταν αρχίζουν τα νέα προγράμματα γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα στην τρέχουσα περίοδο και το λένε κάποια κράτη-μέλη σε εκθέσεις στρατηγικής, ότι επεκτείνοντας την προηγούμενη προγραμματική περίοδο επιβραδύνουμε την ε, υλοποίηση της τωρινής. Αυτό καλό είναι να αποφευθεί. Χρειάζονται πιο πολλές αξιολογήσεις των τρεχών των προγραμμάτων για το μέλλον ε, πρέπει να βελτιώσουμε τη χρήση των δικτών. Οι βασικοί δείκτες είναι σημαντικοί, αλλά δεν χρησιμοποιούνται όπως πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις και αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και στην, τωρινή, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και στην επόμενη. Πιστεύουμε ότι οι αδυναμίες, εις ό,τι αφορά την, τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουμε φαίνεται στην έκθεση στρατηγικής και αυτό ε, αποδεικνύει την ορθότητα των προτάσεων της Κομισιόν για το μέλλον, ιδιαίτερα την ανάγκη εστίασης στο, στα αποτελέσματα, τις επιδόσεις, την σαφή υποβολή εκθέσεων των ε, όσων επετεύθησαν, διαφάνεια, συζήτηση, συζήτηση και για τα αποτελέσματα που επιτεύθηκαν, να μην περιοριζόμαστε στα ασφάλματα και στην απορροφητικότητα, γιατί όπως ε, είπαμε, και όπως λέμε και στην έκθεση στρατηγικής, αυτό είναι κομμάτι της κίνησης προς τη λογοδοσία για τα αποτελέσματα που επετέφθησαν και τους πόρους που δαπανήθηκαν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι προτάσεις μας ως προς αυτό το πλαίσιο για τη μελλοντική πολιτική είναι σωστές και το θετικό είναι ότι υποστηρίχθηκαν και από το Συμβούλιο οι προτάσεις μας αλλά και από εσάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα υπάρχει συμφωνία ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Σταματώ εδώ, υπάρχει πληθώρα υλικού στην ιστοσελίδα μας και μας ενδιαφέρουν οι αντιδράσεις για την έκθεση. Ευχαριστώ. Από ό,τι ξέρω ακόμη δεν θα λάβει το λόγο ο Τζον, οπότε θα μιλήσει μετά όταν έχουμε τις ερωτήσεις που αρχίζουμε τώρα, παρατηρήσεις και υποβολή αλλα αλλά πρώτα-πρώτα η Κωνσταντσα Κρέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πολύ εντυπωσιακή πραγματικά έκθεση για την πολιτική συνοχής και όπως έλαβε χώρα στα κράτη-μέλη μέχρι τώρα, πως υλοποιήθηκε δηλαδή, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και ερωτήσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Κυρίως ε, τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εσείς τονίσατε και ακούγεται εντυπωσιακό ότι δημιουργήθηκαν 400.000 θέσεις εργασίας μόνο τα τελευταία έτη. Αλλά αυτό είναι εντυπωσιακό μέχρι να δει κανείς τα νούμερα ε, των θέσεων εργασίας που χάθηκαν αυξάνοντας την ανεργία αν δούμε δηλαδή συγκριτικά τα στοιχεία δεν κάναμε τίποτα δημιουργώντα 400.000 θέσει εργασία από το Κοινωνικό Ταμείο. Και αν δω τον πίνακα που δείχνει το πού δημιουργήθηκαν αυτέ οι θέσεις εργασία, εκεί η πρώτη είναι η Γερμανία, η οποία από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επλήγει λιγότερο από κάθε άλλη χώρα. Βέβαια, ναι, ε, έχουμε και δημιουργία θέσεων εργασία στην Ιταλία. Αλλά οι άλλες χώρες που συνταράσσονται από την κρίση έχουν μείνει απόξω. Γιατί προφανώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν τα λεφτά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να μετριάσουν την κρίση που τη πλήττει. Και αν συζητάμε τι θα γίνει ε, παραπέρα με το κοινωνικό ταμείο, με τις εγγύσεις για τους νέους, το Youth Guarantee, ε, είναι σημαντικό να μας πείτε πώς μπορούμε ενδεχομένως να καταφέρουμε πιο πολλά πράγματα, να έχουμε πιο πολλές θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Να σκεφτούμε μήπως υπάρχουν κι άλλες μέθοδοι για να στηρίξουμε αποτελεσματικότερα την αγορά εργασίας και Θέλω να μου κάνει κάποια εκτίμηση η Κομισιόν ή να μου δώσει κάποια πληροφορία. Τι προβλέπετε για όλα αυτά. Γιατί για αυτά δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Είναι η Επιτροπή Απασχόλησης υπεύθυνη για το κοινωνικό, αρμόδια για το κοινωνικό ταμείο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε στο μέλλον ούτως ώστε να υποστηριχθούν πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αγορά εργασίας και να επενδύουμε σωστά τα χρήματά μας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρονικό διάστημα που απομένει για να αλλάξουμε ίσως κάποια πράγματα. ή να ενισχύσουμε ή να μην ενισχύσουμε κάποιες πολιτικές που προβλέπονται αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ, Λάμπερτ Βανίστελ Ρόι. Having this report here, wonderful combination with the debate we had. Πάρα πολύ ωραία συνδέεται αυτή η έκθεση με την συζήτηση που έγινε σήμερα το πρωί. Σε σχέση με τις δικές μας επιδόσεις και τις ε, μακροδημοσιονομικές, μακροοικονομικές εξελίξεις. Για πέστε μας. Είναι δυνατόν εμείς εδώ στην Επιτροπή μας να μπορέσουμε εκτός από την πρώτη ματιά που ρίξαμε να κάνουμε ε, σαν και αυτή την έκθεση για το ίδιο θέμα μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Και ίσως μια τέτοια εφαρμοστική έκθεση χρειάζεται, διότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των επιδόσεων χώρων μελών. Οπότε είναι δυνατόν να εμβαθύνουμε στο ίδιο θέμα και να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση σε σχέση με το τι έχουμε πετύχει κατά αυτή την περίοδο και για το τι βελτιώσει μπορούμε να επιφέρουμε για την επόμενη περίοδο. Δεν λέω να γίνει αυτό εδώ και τώρα, ας το σκεφτούμε. Ίσως θα ήταν θετικό. Να εμβαθύνουμε. Α, αυτό δεν ήταν ερώτηση προς την κυρία Γκάφη, λέει Πρόεδρος. Θεωρώ ότι αυτό το λέτε για την συνάντηση των συντονιστών που θα γίνει το απόγευμα. Άλμπριχτ. Έχω δύο παρατηρήσεις, αλλά και δύο ερωτήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό την έκθεση αυτή να την είχαμε λάβει πριν τη σημερινή συνεδρίαση. Είναι ενδιαφέρον θα πρέπει να έχουμε χρόνο όμω δεν έχουμε μελετήσει από πριν. Και μετά να έχουμε ετοιμάσει τι ερωτήσει να τι υποβάλουμε. Αυτό για το μέλλον. Δεύτερη παρατήρηση. Είναι ευχάριστη έκπληξη το πόσε θέσει απασχόληση έχουμε στον Ηνωμένο Βασίλειο λόγω τη νέα ε, πολιτική συνοχή. Τώρα, οι παραμονέ του, Ευρω... του δημοψηφίσματο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, έχουμε και το δημοψήφισμα στη Σκοτία, εκτό ε, μικροφώνου. Δύο ερωτήσει. Η πρώτη αφορά το πολιτισμικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Πέρσι. Το πρόβλημα ήταν ότι τελείωσαν τα χρήματα. Τώρα όμως δεν πιστώνεται ότι πάρα πολλά κρατημέλη δεν είναι έτοιμα. Άρα δεν θα προωθήσουν τα χρήματα. Όμως ακόμα υπάρχουν χρήματα στον προπολογισμό για την πολιτική συνοχή. Άρα, οι πληρωμές είναι τόσο χαμηλά. Οπότε παρά το ότι είναι συγκρατημένες οι δαπάνες, ακόμη λείπουν τα χρήματα. Πολύ σημαντική η ερώτηση αυτή. Γιατί πολλοί συνάδελφοι στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών δεν έχουν υπόψη αυτά τα στοιχεία. Και θεωρούν ότι λόγω της, ε, το ότι δεν είναι προετοιμασμένοι πολλά κρατημένοι μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Όμω βλέπω εδώ ότι ακόμα και με λίγες πλήρωμέ πάλι δεν έχουμε χρήματα. Πολύ σημαντικό. Τώρα για τους δίκτες. Τελευταία ερώτηση. Είχαμε την ε, ευκαιρία να τα συζητήσουμε και ακόμα συζητούμε και στην τελευταία σας ε, διαφάνεια υπήρχε κάτι σε σχέση με τους δείκτες. Μία φράση ημιτελής. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τα δείκτες. Τι είπατε, πώς χρησιμοποιείται, πώς χρησιμοποιείται. Δεν το κατάλαβα γιατί ήταν ε, η μητελής φράση στην διαφάνεια. Είπατε ότι δεν έχει δεν τέτοιου δείκτε. Για πώ έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα τη σημερινή μέρα, λέει η πρόεδρο. Μαρία Ριγκόγεν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στη συνέχεια των όσων είπε ο Γιάννα Αλμπριχτή, έχω και εγώ να παρατηρήσω τα εξή. Είναι χρήσιμη, αναγκαία αυτή η έκθεση, γιατί γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής. Για μένα συνοχή θα πει ανάπτυξη και επενδύσεις. Και επιτρέψτε να έχω κάποιες επιφυλάξεις σε κάποια από τα μέτρα κατά της κρίσης. Αλλά νομίζω ότι αυτά που ακούμε εδώ πέρα είναι καλά μαντάτα. Ότι αυξήθηκαν και τις εργασίες, δημιουργήθηκαν έτσι. Έχουμε την έκθεση του ΩΣΑ που λέει ότι θα πάει η χώρα μου κόντρα στις προβλέψεις, κόντρα στην κρίση σε ανάπτυξη 1,7. Τι λέτε, εν ώψη αυτών των αποτελεσμάτων, των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για να αυξήσουμε την ανάπτυξη σε κάποιες περιφέρειες που την χρειάζονται. Τι θα γίνει με την συγχρηματοδότηση σε σχέση με την χρήση των πόρων. Γιατί έχουμε κάποιες αυτόνομες δικαιωτικές περιφέρειες που έχουν αυτό το θέμα στην ε, Ισπανία. Πρόεδρος. Ο Ήβο θα μας πει ότι όλα τα στοιχεία τα ξέρει των προϋπολογισμών. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς αυτό θα σας πω. Μερικοί από εμάς τα γνωρίζουμε. Αλλά η ερώτησή μου αφορά την Επιτροπή. Αν δείτε το έγγραφο της 16ης Μαΐου, τα στοιχεία σε σχέση με την πολιτική συνολική από τα κράτη-μέλη βλέπετε μόνο το 2013 οι αξιώσει ανέρχονται στα 65 δις δύο φορές περισσότερα από όσα είναι γραμμένο στον προπολογισμό. Και επίσης πριν την πρώτη ενδεκάτου όπου έχουμε τότε 48 δις και μετά τον Νοέμβριο για το 2014 έχουμε 16 δισεκατομμύρια. Είδατε, μας εξήγησετε πώς έχει το τοπίο για τον προγραμματισμό ή τον αναπρογραμματισμό αυτή η αλλαγή των δεσμεύσεων για κάποιες χώρες ονομάζεται επιπρόσθετη δέσμευση. Και βέβαια κάτι το οποίο έχει σχέση με όλα αυτά είναι η ταμιακή ροή που και εδώ πέρα έχουμε προβλήματα. Άρα, σήμερα με το τι ισχύει σήμερα μπορεί να έχουμε κάποιες δεσμεύσεις μέχρι το 2017. Δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει θέμα στο αποθεματικό και οι χώρες που είναι στο 82% του ΕΠ ε, βλέπουμε ότι ε, δεν κατατείνουν όλα αυτά τόσο αλληλένδετα στο να βρεθεί διέξοδος εύκολα. Θα πρέπει η Γενική Διεύθυνση για τα Δημοσιονομικά και τον Προπολισμό να συνεργαστεί με την ε, Γενική για τα Περιφερειακά που δεν έχει συνθεί μέχρι τώρα. Πεςτε μας δύο λόγια πάντως για το πού, σε ποιους τομείς γίνεται αυτός ο αναπρογραμματισμός, σε ποιες χώρες, σε ποιο τομέα και κυρίως τι είδους αναπρογραμματισμός είναι αυτός. Γιατί κάποιες χώρες αν σε αυτή την περίοδο προχωρήσουν προς κάποιο είδους συμφωνία για διαχείριση των επενδύσεων, τότε θα δούμε αν γίνεται να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που να βοηθά στην επίτευξη των στόχων. Γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοια επικάλυψη των φάσεων που να μην μπορεί να αρχίσει όταν πρέπει η κάθε φάση το κάθε πρόγραμμα. Αν μπορείτε Δώστε μας κάποια στοιχεία, κάποια αποτελέσματα για τον επαναπρογραμματισμό. Γιατί όταν φτάσουμε στην επόμενη περίοδο επταετίας προγραμματισμού θα πρέπει να τα κράτη-μέλη να έχουν ε, αυτά τα στοιχεία διάθεσή τους. Πρόεδρος, δεν βλέπουμε να ζητεί κανείς το λόγο, οπότε θα δώσω κύριε Γκάφη και πάλι το λόγο. Θα κάνω ό,τι μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ που τις υποβάλλατε. Συγγνώμη αν κάτι παραλείψω. Πάντα το θέμα είναι τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας. Όλοι γι' αυτό ενδιαφέρονται. Και αυτό και έχουμε αυτούς τους ε, εμπειρογνώμονες, αξιολογητές, οι οποίοι κάθε χρόνο κάνουν αυτόν τον υπολογισμό, καταλαβαίνουν, ξέρουν τι γίνεται. Οπότε και έτσι αυτή η σχετική έκθεση σε κάνα δύο μήνες θα είναι έτοιμη για να τη μελετήσετε. Αναφέρονται λοιπόν αυτά τα στοιχεία στο τι μας λένε τα κρατημέλη για αυτές τις εργασίες. Να δείτε ότι έχουμε εξέλιξη του σύστηματος των δικτών. Καταρχήν είναι σε χαλαρό επίπεδο οι δείκτες κατά την προγραμματισμό. Και ο σκόπος είναι να έχουμε ποσοτικούς δείκτες, όπου γίνεται μας ζήτησε ο Γενικός Διευθυντής να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και είπαμε στα κρατημέλια παρακαλώ γίνεται να κάνετε μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσετε λίγους δείκτες ούτως ώστε να είναι κάτι που να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν κάτι σε συμφωνία κυρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Πάντως πρόκειται για πιλωτική πρωτοπόρα προσπάθεια. Γι' αυτό και είμαι επιφυλακτική όσον αφορά αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει όλοι να έχουν τα ίδια μέτρα όταν έχουμε την ε, συλλογή των, ε, των δικτών και τα, τα αθρηστικά τέλος πάντων. Αλλιώς νοθεύεται. ο υπολογισμό. Πολλέ φορέ, α πούμε κάποιοι παλιούν κάποια μηδενικά, μπερδεύουν τα, τα, τα, δεκαδικά και όσον αφορά τώρα τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, υπάρχει μια χρονική υστέρηση. Αυτά τα δεδομένα ανατρέχουν στο 2011. Και τα στοιχεία για θέσει εργασία συνήθω τα έχουμε όταν ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα. υπάρχει κάποια Και είναι ατελή τα δεδομένα γιατί κάποια κρατημέλη τα χρησιμοποιούν, κάποιοι άλλοι κάνουν λάθος κωδικοποίηση και επίσης πολλές φορές δεν περιέχονται οι θέσεις εργασίας που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Κοινωνικό Ταμείο υπολογίζει τα χαρακτηριστικά των ε, ε, απασχολουμένων και τι γίνεται μετά την κατάρτισή τους. Και έτσι όμως βοηθούνται οι επιχειρήσεις όσον αφορά την έρευνα και την καιροδομία. Οπότε, γι' αυτό μπορούμε να δούμε τι θα γίνει με τα δεδομένα κατά αυτή την περίοδο. Κύριε Βαγνίστερ είχατε ψήφισμα με βάση τη δική μας τελευταία, η προηγούμενη στρατηγική έκθεση. ...18 Τετάρτου την εγκρίναμε. Άρα ισχύει εδώ και αρκετό καιρό. Και όποτε θέλετε να, να την ξανασυζητήσουμε. Τώρα για την έλλειψη χρημάτων στον προπολογισμό. Εύστοχα αυτά που είπατε. Όντως υπάρχει πρόβλημα. Αν δηλαδή τα κατημερινή διαλέξουν να απορροφήσουν αυτά τα οποία τους έχουν ε, καθορίσει, τότε θα υπάρξει τις επόμενες χρονιές αντίστοιχη δέσμευση κονδυλίων στον προπολογισμό. Έχουμε πάντως 55% των πόρων που θα πρέπει να απορροφήσουμε μέχρι το 2015. Όχι, συγγνώμη, λέει ο 55% των πόρων για το οποίο θα πρέπει να υπάρχουν ε, αξιώσεις καταβολής. Πολλές φορές υπάρχει καθυστέρηση σε σχέση με την υποβολή αυτών των αξιώσεων. Αυτό τώρα για τις πληρωμές. Όσον αφορά τώρα τις πληρωμές και υποχρεώσεις, βασικά ο αναπρογραμματισμός έχει σχέση με τις δεσμεύσεις, τις υποχρεώσεις. Όχι με τις πληρωμές. Παρ' όλα αυτά, στη στατική έκθεση λέμε ποιε είναι οι επιφυλάξεις μα, λέμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές καθυστερήσει σε πολλούς τομείς και επίσης βλέπουμε να υπάρχει, το υπάρχει σε κάποιους άλλους τομείς. Και έρχονται τα κράτη-μέλη. Το 2014 ή ακόμα και το 2015 και ζητούν αναπρογραμματισμό σε κάποιους τομείς όπου είναι κορεσμένοι. Το θέμα είναι κατά πόσο θα το κάνουμε αυτό. Και η στρατηγική έκθεση τι λέει, ότι κάποιοι κρατημέλοι ίσω θέλουν να κάνουν αναπρογραμματισμό το 2014-2015 σε κάποιου τομεί όπου είναι ευκολότερο να, να δαπανηθούν χρήματα όπω τοπικοί δρόμοι. Και εμεί είπαμε ότι οποιοδήποτε ε, παραπάνω αναπρογραμματισμό θα πρέπει να αφορά κάποιε επενδύσει που είναι ε, που μεγιστοποιούν την ε, την αποτελεσματικότητα των πάντων και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Όλα αυτά θα θέτουμε επί της τραπέζης για συζήτηση με εσά, με τα κράτη-μέλη, με το Συμβούλιο και έτσι να μπορούμε να έχουμε διαφάνεια για να διαπιστώσουμε το ποια θα είναι η επόμενη κίνηση και ποιοι είναι οι κίνηση. Τώρα επίσης για τον προγραμματισμό, αν θέλετε λεπτομέρειες υπάρχουν. Έχουμε στοιχεία, μερικά από τα οποία είναι στο 7.3 και 7.4, τους πίνακες αυτούς, σελίδες 54 και 55 στο στο έγγραφο εργασία για το προσωπικό. Ελπίζω σας απάντησα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν περαιτέρω σχόλια. Ε, καθίσταται σαφές ότι αυτό που μας ενδιαφέρουν είναι τα αιτήματα καταβολής ε, πληρωμών κατά το, τη νέα οικονομική περίοδο. Εάν λοιπόν ε, δεν ε, καθυστερήσουμε ε, εάν λοιπόν καθυστερήσουμε θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Πρέπει να μην καθυστερήσουμε, δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται η ιστορία ως προς την αρνητική της πτυχή. Δεν ξέρω κατά πόσο, Τζον, θέλεις κάτι να προσθέσεις, ναι. Ο Τζον Βόλες, μια και είμαι εδώ. Ευχαριστώ. Ως προς την απασχόληση, δύο διασαφήσεις. Η Βερόνικα μίλησε για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης από ΜΜΕ, καινοτομίας και έρευνας. Άρα ανακύπτει και το ερώτημα της κυρίας Κρέλ. Υπό την πολιτική συνοχής υπάρχουν αιτήματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Από, πλε, από πλευράς λοιπόν υποδομής δημιουργούμε ε, θέσεις εργασίας όπως στον τομέα των κατασκευών, αλλά δεν πρόκειται για βιώσιμες θέσεις εργασίας, μόνιμες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό δεν πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή τη θριαλίδα ότι δηλαδή υπάρχουν ή δημιουργούνται μόνιμες θέσεις εργασίας, άρα αυτές δεν τις ε, προσμετρούμε. Έχετε ε, δίκιο όταν μιλάτε για την ε, κλίμακα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με την κλίμακα απώλειας θέσεων εργασίας. Άρα η πολιτική συνοχής δεν στοχοθετείται ε, άμεσα ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Γι' αυτό έχει σημασία τα κράτη-μέλη πού θα επενδύσουν, διότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι θέμα ύψης της σημασίας όπως και το 2006 όταν συζητήθηκε ως προς τον επαναπρογραμματισμό. Ε, έτσι έχουν τα πράγματα όπως είπατε και εσείς. Μιλάμε για θεματικό επαναπρογραμματισμό έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε σχέση με το πώς είχαν ε, οριστεί ε, αρχικά, δηλαδή περνάμε από το δικό δίκτυο στο σιδηροδρομικό ή στο διατροπικό. Υπάρχουν αλλαγές μεταξύ προγραμμάτων και υπάρχουν και κινήσεις ε, στα κράτη-μέλη ως προς τη χρήση των κονδυλίων. Δηλαδή, ορισμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης πέρασαν στο ΕΚΤ. Όπως είπε και η συνάδελφος, η κυρία Γκάφη, έχουν γίνει αλλαγές χρήσης ο νέος επαναπρογραμματισμός θα είναι αποδοτικός γιατί ε, δεν έχουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως προς την ε, ε, νέα κατανομή. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να γίνονται μεγαλύτερες αλλαγές όσο προχωρούμε στο πρόγραμμα αυτό το θέμα της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, πού πρέπει να επενδύσουμε, αυτό είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας στην ατζέντα μας. Έχουν γίνει έρευνες, αλλά δεν έχουμε καμία σιγουριά για το πού θα πρέπει να επενδύσουμε για να φτάσουμε σε ανάπτυξη και απασχόληση. Υψηλότερους δείκτες δηλαδή. Ποιο θα έρθει πρώτο, η ανάπτυξη ή η απασχόληση. Γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη δημιουργεί απασχόληση αλλά τι δημιουργεί ανάπτυξη. Εδώ υπάρχουν προκλήσεις και δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Θα θέλαμε να συζητηθεί το θέμα με ακαδημαϊκούς κύκλους για να φτάσουμε σε μεγαλύτερη, μεγαλύτερη συνένεση γιατί έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον. Η Κωνσταντσα Κρέλ. Αυτό σημαίνει ότι τη η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. From the ESF. And you don't have... Οι 400.000 θέσεις εργασίας ε, σημαίνει ότι έχετε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με τα 15 εκατομμύρια που έχουν αποδοθεί. Αυτό τι σημαίνει. Ε, έχετε στατιστικά στοιχεία για αυτούς που απασχολήθηκαν, δεν απασχολούνται πλέον και μπορούν να ξαναενταχθούν στην αγορά εργασίας. Γκάφη. Οι αξιολογήσεις του ΕΚΤ δείχνουν ότι έχουμε 12,5 συμμετέχοντες στο ΕΚΤ γιατί τα 15 εκατομμύρια φορούν κάθε τύπο κατάρτισης και η αξιολόγηση δείχνει ότι 2,4 ε, εκατομμύρια βρήκαν ε, θέση εργασίας μετά από εξάμηνη μαθητεία από τα 12,5 εκατομμύρια. Αυτό ήταν πολύ θετικό, αλλά δεν, μπορεί, δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια με αυτά τα 4 εκατομμύρια ε, που θα πρέπει να βρουν θέσεις εργασίας μέσω των 400.000 θέσεων. Χρειαζόμαστε ε, περισσότερα στοιχεία για να δούμε, να τα διερευνήσουμε αυτά τα στοιχεία, να ξέρουμε επακριβώς τι έχει συμβεί. Ήβο, ποια είναι η θέση σας, η Επιτροπή προβάλλει προτάσεις αύξησης της συμμετοχής του Κοινωνικού Ταμείου Μιλάμε για ένα 25% τουλάχιστον. Σύμφωνα με τις δικές σας έρευνες, αυτή είναι σωστή προσέγγιση ή όχι. Δεν το έθεσα πολύ ε, διπλωματικά. Η μόνη εξήγηση είναι, είναι ότι εμείς δείξαμε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή το μερίδιο του ΕΚΤ θα είναι μεγαλύτερο και άρα θα έχουμε και περισσότερες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά επειδή δούλεψα για το ΕΚΤ Πιστεύω ότι οι δεξιότητες αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ε, πρόθεση της ανάπτυξης. Αυτή είναι η θέση της ε, Επιτροπής. Yes, we Προς το συνάδελφο Γκουντμάνης Εκτός μικροφώνου η παρέμβαση. Για την Πολωνία έχετε δημοσιεύσει, έχει δημοσιευθεί μία έρευνα για το πού θα πρέπει να διατεθούν τα ευρωπαϊκά ε, κονδύλια. Και στην Πολωνία ε, λένε όλοι οι συμμετέχοντες ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για την εκπαίδευση. Αυτό λέει η πλειοψηφία. Στην Πολωνία ποτέ δεν λέμε αυτά που σκεφτόμαστε, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι έγινε κάτι τέτοιο. Ιωακίμ, ξέρουμε εκ πείρας ότι χρειάζεται μία ε, παρέμβαση με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε. Εάν δημιουργούνται τεχνητά θέσεις εργασίας μέσω ΕΚΤ, τότε ε, αυτό το πλαίσιο δεν είναι καθόλου αποδοτικό. Αυτό το είχαμε δει και στην πρώην Ανατολική Γερμανία και στο Βερολίνο. Ε, θέλουμε τα ε, πρόσωπα να μην υπάρχουν στις λίστες του ΟΑΕΔ και πολλές φορές ε, χρησιμοποιούμε με τεχνητά, μέσα για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, κάτι το οποίο είναι πολύ ε, λανθασμένο. Γιατί αυτά τα φυσικά πρόσωπα ξαναβρίσκονταν εκ νέου στη, στην ανεργία και μετά έμπαιναν στα στατιστικά στοιχεία ανεργίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε το προφίλ των μέτρων στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διατηρήσιμη απασχόληση είναι ο στόχος, γιατί και η κατάρτιση και η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση ε, εκεί αποσκοπεί. Ε, όσο υπήρχε χρηματοδότηση βέβαια όλα αυτά λειτουργούσαν καλύτερα. Όταν έλειψε η χρηματοδότηση δεν μπορούσαν πια οι επιχειρήσεις να έχουν αυτούς τους ε, καταρτιζόμενους και κατήγγυλαν τις συμβάσεις. Και γίνεται αυτό, μην έχουμε αυταπάτες. Οπότε τέτοια μέτρα δημιουργίας απασχόλησης χρειάζονται εκεί που υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει να χρηματοδοτείτε. Αλλά τώρα όταν ε, Λέμε ότι 52% των διαρθρωτικών ταμείων ε, είναι ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, εκεί υπάρχει πρόβλημα γιατί μιλάμε για τις πιο αναπτυγμένες χώρες. Στην Πολωνία αναφέρθηκε ότι η κατάρτιση είναι το πιο σημαντικό, εκπαίδευση-κατάρτιση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα προσόντα, στην εξειδίκευση και να μπαίνει κανείς με καλύτερη εξειδίκευση και πιο πολλά προσόντα στην αγορά εργασίας. Βέβαια δεν γίνεται η εξειδίκευση ως αυτός σκοπός. Γιατί στο Βερολίνο τη δεκαετία του 90 εξειδικεύτηκαν πάρα πολύ σε συγκεκριμένες ειδικότητε που δεν χρειαζόντουσαν στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε. γιατί πολλές φορές και τα στατιστικά στοιχεία υπολείπονται της πραγματικότητας. Απασχόληση δημιουργείται μόνο μέσα από, βιώσ, από διατηρήσιμα μέτρα για να είναι και διατηρήσιμη η απασχόληση. Και εκεί ε, πρέπει να δώσουμε έμφαση, να υπάρχει δηλαδή μια, μονι, μια μονιμότητα. Είναι σημαντικό επίσης οι επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα χρέωσης γιατί δεν τους βοηθάνε οι τράπεζες ε, αυτές οι επιχειρήσεις, κατά τα άλλα, πολλές φορές είναι καθόλου υγιείς και παραγωγικές. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να υποστηριχθούν, βεβαίως. Όχι όμως με μέτρα τεχνητά που δεν βοηθούν τους εργαζομένους, γιατί αυτά τα μέτρα μόνο ε, μικρό αποτέλεσμα, μικρής διάρκειας αποτέλεσμα έχουν, βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Η Κομισιόν θέλει να μας πει, να απαντήσει. Θα απαντήσει, ε, ε, ε, αλλά εδώ πρέπει να διακόψουμε και ευχαριστώ όλους.